Good morning, uh, everyone. Uh, my name is Richard Czarnecki. Χαίρετε. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Σαρνέτσκι από την Πολωνία, Ευρωβουλευτής. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε στη δεύτερη αυτή ημέρα μιας πολύ σημαντικής διακοινοβουλευτικής διάσκεψης ε, για την πολιτική ασύλου και μετανάστευση Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνέπειες για τη ε, κοινοβούλια των ε, χωρών της διεύρυνσης. Χαίρομαι ιδιαίτερως που βλέπω εδώ τους συναδέλφους μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα που θα μας απασχολήσει και σήμερα, όπως γνωρίζουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει άνευ προηγουμένου κρίση. Η μετανάστευση είναι ε, πρώτη προτεραιότητα στο πολιτικό θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζει άμεσα τις ε, χώρες ε, των Δυτικών Βαλκανίων και ιδιαίτερο στην πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και τη Σερβία. Χώρες οι οποίες έχουν δράσει ως υπεύθυνοι εταίροι στη διαχείριση των ροών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται λοιπόν με την ε, ανάπτυξη των ε, μέσων και των, ε, του δυναμικού για την αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων και την καταπολέμηση της λαθρεάς διακίνησης ατόμων. Η Τουρκία, από την άλλη, έχει υποδεχθεί δύο εκατομμύρια σύρων προσφύγων και είναι η, χώρα που, ανα, που υποδέχεται το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων στον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξακολουθήσει να επιδεικνύει αλληλεγγύη η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας ε, επιδεικνύει ήδη επιτυχίες πιστεύω. Οι ροές μεταναστών από την Βαλκανική Οδό έχουν ουσιαστικά πάυσει. Η δέσμευση της Τουρκίας και για την υλοποίηση της ελληνοτουρκικής διμερούς συμφωνίας επανεισδοχής ε, φαίνεται να προχωρεί και αυτή σε ε, καλή εφαρμογή. Ένα κοινό σχέδιο δράσεως λοιπόν θα μπορούσε από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσφέρει και ε, στην, ε, στους Σύρους που βρίσκονται στην Τουρκία ικανοποιητική προστασία. Πρέπει επίσης να συζητήσουμε το θέμα του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να υπάρξει ορθή διαχείριση και προστασία των εξωτερικών συνόρων έτσι ώστε να υπάρχει διάκριση μεταξύ προσφύγων, εκείνων δηλαδή που δικαιούνται είσοδο, και εκείνων που δεν δικαιούνται. Τα θαλάσσια σύνορα ωστόσο δεν είναι ευχεροί στην, στον έλεγχο, δεν είναι πρόσφορα σε έλεγχο. Θα γνωρίζετε ασφαλώς το γεγονός αυτό, το έχουμε ξανασυζητήσει. Και θα ήθελα ακόμη να συμπληρώσω ένα μήνυμα. ότι η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη διαδικασία της διεύνησης και τη μετανάστευση θα πρέπει να κοιτάει προς τα μπρος και να είναι να προλαβαίνει τις κρίσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά της, ε, την αυλή της, τον την εγγύ της γειτονία, δηλαδή τα Δυτικά Βαλκάνια. Έχουμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα συζητήσεων διαφόρων θεμάτων σήμερα, με θέματα που συμπεριλαμβάνουν την παρουσίαση της κατάστασης στα ευρωπαϊκά σύνορα προς τις χώρες διεύρυνσης, σε σχέση με τη μεταναστευτική κρίση, ενίσχυση των λειτουργικών ε, δυνατοτήτων, δράση της εκτελεστικής εξουσίας, κοινοβούλια ε, και χάραξη πολιτικής, ώστε και η εκτελεστική ε, εξουσία αλλά και η κοινωνία των πολιτών να συνεργάζονται, διακοινοβουλευτική συνεργασία και περιφερειακή συνεργασία των αρμοδίων αρχών θα είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν. Τα θέματα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι θέματα κυρίως της Επιτροπής των Εξωτερικών Υποθέσεων, Επιτροπής ΑΦΕΤ, όπως τη λέμε. Είναι θέματα λοιπόν τη Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, η οποία είναι μεταξύ των συνδιοργανωτών της ε, παρούσας διάσκεψης. Και όπως γνωρίζετε, είναι μία εκ των πρωταγωνιστών του σχεδιασμού και της υλοποίησης εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η ΑΦΕΤ αποφασίζει την διάθεση των κονδυλίων τον τρόπο με τον οποίο θα διατίθεται δηλαδή, τα κονδύλια για την υλοποίηση εξωτερική πολιτική και των αξιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και επιβλέπει τη διαδικασία διεύρυνση. Σα ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σα εδώ. Προσβλέπουμε σε μια δεύτερη μέρα επικοδομητικών και ενδιαφερουσών συζητήσεων. Περνάει γρήγορα ο χρόνος και έτσι δεν θέλω να καθυστερήσω περισσότερο. Θα σας παρουσιάσω τους ομιλητές μας για σήμερα. Έχω την χαρά και τιμή να καλέσω τον εκτελεστικό διευθυντή της Frontex, κύριο, τον κύριο Φαμπρίς Λεζουρί, να πάρει το λόγο για τα θέματα της μετανάστευσης και των κρίσεων σε σχέση με τα ευρωπαϊκά σύνορα με τις χώρες σας, προς τις χώρες σας. Ο κύριος Λεσρή είναι γαλλικής καταγωγής. Έχει εργαστεί στο Υπουργείο Ιστορικών της Γαλλίας και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορα θέματα σχετικά με τη Συμφωνία Σέγγεν, τη μετανάστευση και το διεθνές δίκαιο. Η Frontex πρόσφατα δημοσίευσε την ανάλυση κινδύνου για τα Δυτικά Βαλκάνια. Ως εκ ο κύριος Λεζουρή θα μπορούσε ίσως να μας ενημερώσει λεπτομερέστερα για το θέμα αυτό στη διάρκεια της παρουσίασής του. Η έδρα της Frontex βρίσκεται στην πατρίδα μου, την Πολωνία. Και εύχομαι τα καλύτερα και για τη Frontex και για τις λοιπές σχετικές ε, υπηρεσίες. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Ε, ε, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσουμε κάποια αριθμητικά στοιχεία και τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τις ε, παράτυπες διελεύσεις εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και θα ήθελα να σας πω ορισμένα πράγματα σε σχέση με την συνεργασία της Frontex με τις χώρες τις οποίες εκπροσωπείται σήμερα εδώ. Οπότε καταρχάς θα ήθελα να ξεκινήσω με την συνολική κατάσταση στα εξωτερικά ε, σύνορα. Από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο η Frontex έχει καταγράψει 330.000 παράτυπες διελεύσεις σύνορων ε, στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Αυτό είναι δύο φορές μεγαλύτερο από την ίδια περίοδο την αντίστοιχη του 2015, αλλά, και αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη, τον Απρίλιο, και αυτό και πάλι επιβεβαιώθηκε το Μάιο του τρέχοντος έτους ε, η, αιτή, ε, η, η αιτήσια παράτυπη διέλευση που καταγράφηκε εκείνο το μήνα ήταν χαμηλότερη από την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή την άνοιξη του 2016 βλέπουμε μία ε, σημαντική μείωση παράτυπων διελεύσεων ε, των, συνόρων της, των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Θα ήθελα επίσης ε, να σας πω ότι τη στιγμή που ε, μιλούμε, ο αριθμός των μεταναστών που περνούν από τη Λιβύη ή από την Αίγυπτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ υψηλότερος από τον αριθμό των παράτυπων μεταναστών που, προέρχονται, που, από, που περνούν από την Ελλάδα ή από την Τουρκία. Δηλαδή, η Frontex το Μάιο κατάγραψε κατέγραψε 17.000 μετανάστες προερχόμενους ε, μέσω της κεντρικής Μεσογείου, μέσω της Ιταλίας στην Ευρώπη και τον Μάιο καταγράψαμε λιγότερο από 1.500 μετανάστες ε, που πέρασαν στην Ένωση μέσω των ελληνικών ε, νησιών και της Τουρκίας. Αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη και έχει σημασία για τη σημερινή συζήτηση μαζί σας. Αν συγκρίνω τα νούμερα και εστιάσω στην, ε, ανατολική, την, στην οδό της Ανατολικής Μεσογείου, το Μάιο, όπως είπα, καταγράψαμε περίπου 1.500-1.800 ε, μετανάστες, 4.300 ε, είχαμε τον Απρίλιο που πέρασαν από την Τουρκία ε, στην Ελλάδα και απλώς για να συγκρίνω, το Μάιο του 2015 η Frontex είχε καταγράψει 20.000 παράτυπους μετανάστες που πέρασαν από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά. Πέρσι λοιπόν το Μάιο 20.000 από την Τουρκία πέρασαν στα ελληνικά νησιά. Φέτος την ίδια περίοδο περίπου 1.500 άτομα πέρασαν από την Ελλάδα, από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 50-60 άτομα κατά μέσο όρο που ε, περνούν στην Ευρώπη, κάτι το οποίο βέβαια καθιστά ευκολότερη την κατάσταση σε σχέση με, το, με την ε, προηγούμενη χρονιά. Θα ήθελα τώρα να περάσω στην ε, οδό των Δυτικών Βαλκανίων ε, που είναι άμεσα ε, συνδεδεμένη με την οδό της Ανατολικής Μεσογείου αλλά τα αριθμητικά στοιχεία επίσης καταδεικνύουν μείωση. Δηλαδή τώρα μεταξύ Κροατίας και Σερβίας η Κροατία δεν έχει αναφέρει παράτυπη διέλευση συνόρων τον Μάιο. Ε, ίσως υπάρχει μια καθυστέρηση στις στατιστικές, αλλά σε κάθε περίπτωση το Μάρτιο είχε αναφέρει 1.700 ανθρώπους, ε, παράτυπους μετανάστες, ε, που ε, πέρασαν από τη Σερβία και τον Απρίλιο ήταν ακόμη λιγότεροι και τώρα πλέον έχει σχεδόν εξαφανιστεί αυτή η οδός, δεν χρησιμοποιείται πλέον. Πρέπει να τονιστεί ότι στο σύνορο μεταξύ Σερβίας και Ουγγαρίας υπάρχει αύξηση παράτυπης διέλευσης συνόρων από τη Σερβία στην Ουγγαρία. Το Μάιο εντοπίσαμε πάνω από 3.200 μετανάστες που πέρασαν από τη Σερβία στην Ουγγαρία αν προσπαθήσουμε λοιπόν να κατανοήσουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα Δυτικά Βαλκάνια και τι ακριβώς συμβαίνει ε, μεταξύ της Ελλάδας, των Δυτικών Βαλκανίων και των κρατών μελών της Ένωσης στην Κεντρική Ευρώπη, μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ότι στην Τουρκία μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει σαφής παρακολούθηση για διαφορετικούς ε, λόγους. Ε, υπάρχει αυτή η δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας ε, που έγινε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το υψηλότερο επίπεδο ηγετών από πλευράς Τουρκίας. Αυτό είναι σημαντικό βήμα στη συνεργασία είναι σημαντικό βήμα όταν βλέπει κανείς ότι οι δραστηριότητες παρακολούθησης Μπορούν να προχωρήσουν, υπάρχουν διαδικασίες ε, ακτοφυλακής, ε, ε, εποπτείας, αλλά και εσωτερικές στην Τουρκία για την καταπολέμηση των λαθροδιακινητών. Υπάρχει ακόμη ένας παράγων που είναι ο έλεγχος που διεξάγεται από την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στα χερσαία σύνορα της Μακεδονίας. Αυτοί οι δύο παράγοντες λοιπόν, μαζί με τη δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, εξηγούν το φαινόμενο ότι τώρα δηλαδή αυτή η οδός της Ανατολικής Μεσογείου και των Δυτικών Βαλκανίων, οι δύο οδοί, είναι κλειστές θα έλεγα, ούτως πύλη, συγκρινώντας με τα αριθμητικά τα σχετικά. Υπάρχει ένας άλλος παράγων. Η ανάπτυξη, ίσως να ισχύει, ε, κάποιων σκαφών του ΝΑΤΟ, με τις συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Άρα έχουμε πιο πολλές ε, περιπόλους στις ε, τουρκικές ακτές. όπως βλέπετε ένα σύνολο παραγόντων οδηγεί στο φαινόμενο αυτό, στο γεγονός δηλαδή ότι έχει τεθεί υπό έλεγχον αυτή η οδός της μετανάστευσης. Ωστόσο πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι υπάρχουν χιλιάδες μεταναστών αποκλεισμένοι τώρα στην Ελλάδα, στην υπηρετική χώρα, σημειώνω. Θα θυμάστε ίσως ότι οι ελληνικές αρχές άρχισαν την, επανεγκατα... την επανεγκατάσταση μεταναστών, με την κατάσταση επαναστών από την Ιδωμένη. Ε, μετακινήθηκαν λοιπόν από την Ιδωμένη προς άλλες τοποθεσίες αυτοί οι μετανάστες, άλλες περιοχές της υπηρετικής χώρας. Πρόκειται για 13 περίπου χιλιάδες μετανάστες που βρίσκονται στην ελληνική πλευρά των χερσαίων συνόρων, οι οποίοι μετανάστες ενδέχεται να αποπειραθούν να ε, αντιπαρέλθουν τους ε, συνοριακούς ελέγχους, είτε για να ε, περάσουν στην πρώην Δημοκρατία της Μακεδονίας, είτε να προσπαθήσουν να αντιπαρέλθουν τους βουλγαρικούς, ελληνοβουλγαρικούς συνοριακούς ελέγχους ή αντίστοιχα της Αλβανίας, τα σύνορα. Πάντως, είναι πολύ περιορισμένη αυτή η αριθμή των μεταναστών. Το οξύμορο στην υπόθεση είναι ότι τα σύνορα αυτά τώρα έχουν τεθεί υπό έλεγχο η διάγνωση εναλλακτικών είναι η ανακάλυψη εναλλακτικών οδών ίσως είναι πιο δύσκολη και τελικά ίσως η κατάληξη είναι ότι εκείνοι που έχουν αποκλειστεί στην Ελλάδα ή και στην Τουρκία αντίστοιχα μετανάστες που θα ήθελαν να ε, περάσουν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ίσως αναζητήσουν εναλλακτικέ οδούς και ίσως αυτό οδηγήσει και σε ε, κατακαιρματισμό των ε, ροών. Δηλαδή, ίσω χωριστούν σε διαφορετικέ ομάδε με ροέ ε, από την Ελλάδα στην Αλβανία, από την Ελλάδα στην Βουλγαρία, στην πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία. Αλλά ενδεχομένω, όπω είδαμε ήδη, και απευθεία διαθαλάσσει από την Ελλάδα προς την Ιταλία ή απευθεία πάλι διαθαλάσσης από Τουρκία προς Ιταλία απευθείας ή, και αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερος γιατί είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η οδός, από την Αίγυπτο διαθαλάσσης προς την Ιταλία. Έχουμε διαπιστώσει αύξηση αφήξεων απευθείας από την Αίγυπτο στην Ιταλία. Κάθε χρόνο την Άνοιξη υπάρχει αυτή το φαινόμενο. Ε, ωστόσο, πρέπει να το κοιτάξουμε για φέτος και με δεδομένο το κλείσιμο της Ανατολικής Οδού των Βαλκανίων και επίσης σε σχέση με τις επιλογές που θα μπορούσαν να έχουν μετανάστες που επιλέγουν ε, την ε, ε, λύση αυτή από την Αίγυπτο διαθελά στην Ιταλία. Δηλαδή είναι απλώς μια μετακίνηση ροών από την Τουρκία προς την Αίγυπτο ή πρόκειται για μετακίνηση ροών από τη Λιβύη στην Αίγυπτο. Πρέπει αυτό να το παρακολουθήσουμε λοιπόν στενά. Αλλά ο κύριος κίνδυνος είναι ότι μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των θυμάτων. Γιατί το ταξίδι διαθαλάσσης από την Αίγυπτο στην Ιταλία είναι μακρύ και τα εγκληματικά δίκτυα είναι ε, αμήλικτα. Οι συνθήκες ε, του ταξιδιού είναι πολύ σκληρές για τους μετανάστες. Και τώρα επιτρέψτε μου να σας δώσω μια επισκόπηση για το καλοκαίρι του 2016. Ίσως η εστίαση τώρα να γυρίσει προς τις ε, οδούς της κεντρικής Μεσογείου, δηλαδή ίσως να αφορά λιγότερο τις χώρες σας, εσάς που εκπροσωπήσετε εδώ, στην αίθουσα αυτή, αυτή η εξέλιξη, αλλά έπρεπε να το επισημάνω, οφείλω να το επισημάνω, σε σχέση με την Ανατολική Μεσόγειο. Διαπιστώνουμε ότι πολλοί μετανάστες από τη Συρία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν αναμένουν στην Τουρκία και ξέρουμε ότι εάν οι διάφοροι εμπλεκόμενοι φορείς ε, που ασχολείται με την υλοποίηση της δήλωσης, κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, εντατικοποιήσουν τις περιπόλους, μάλλον ε, χαλαρώσουν τις περιπόλους που τώρα είναι εντατικές, αυτό θα οδηγήσει και σε διαφορετικές εξελίξεις ως προς τις ροές. Αυτά για την παράτυπη διέλευση των συνόρων. Τώρα θα ήθελα να πω Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ελλάδα. 57.000 μετανάστες έχουν μείνει αποκλεισμένοι στην Ελλάδα. Ε, μετά τη δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, μετά την 20η Μαρτίου δηλαδή. Οι περισσότεροι μετανάστες που καταφτάνουν στα ελληνικά νησιά προερχόμενοι από Τουρκία καταθέτουν αίτηση ασύλου όπως γνωρίζετε, ε, μέρος της δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας αφορούσε συμφωνία για επανεισδοχή από την Ελλάδα στην Τουρκία. Η Frontex προσφέρει την υποστήριξή της στις ελληνικές αρχές σε αυτή τη διαδικασία της επανεισδοχής. από τις αρχές Απριλίου η Frontex έχει υποστηρίξει τις επιχειρήσεις επανεισδοχής. Λιγότεροι από 500 μετανάστες ήταν ε, ε, αυτοί οι οποίοι επαναπροωθήθηκαν από την Ελλάδα στην Τουρκία. Σε συνεργασία με την Ελλάδα οργανώσαμε διαθαλάσσεις την επιστροφή αυτών των ανθρώπων ε, με τα φεριμπότ, αλλά και αεροπορικός από τα ελληνικά νησιά στα άδανα της Τουρκίας. Η πρόκληση λοιπόν τώρα για τις ελληνικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να παραμένει ο αριθμός των επανειστοχών σχετικά χαμηλός επειδή ε, βρίσκεται σε στενοπό ένα κομμάτι της διαδικασίας της ε, διεκπαιρέωσης των αιτήσεων ασύλου στην Ελλάδα, παρά την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν συμφορήσεις, είναι τεράστιο το έργο για τις αρχές που έχουν επιφορτιστεί με το άσυλο, με την διεκπαιρέωση των αιτήσεων, μια-δυο αποφάσεις του εφετείου ή μάλλον Επιτροπής Προσφυγών στην Ελλάδα και εφετείων της Ελλάδας που είπαν ότι θεωρούν πως για ορισμένους πρόσφυγες η Τουρκία δεν είναι ασφαλής χώρα, τουλάχιστον έτσι εκτιμούν αυτοί ε, οι δικαστικές αρχές. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν και θέλω να καταστήσω σαφές πως η Frontex επαναπροωθεί μετανάστες μόνο των οποίων οι αιτήσει ασύλου δεν εκκρεμούν. Αυτό σημαίνει πως δεν ασχολούμαστε, γιατί δεν είναι στην εντολή μας, δεν ασχολούμαστε με την αξιολόγηση της αιτήσεως. Πάντως βεβαιωνόμαστε πάντα για την επαναπρόθεση ότι δεν εκρεμεί αίτηση ασύλου στην Ελλάδα και ότι με, σε νομικούς όρους, ε, ότι νομικά δεν υπάρχει κόλλημα για την επαναπρόθεση του ατόμου αυτού στην Τουρκία. η πρόκληση σε σχέση με τις διαδικασίες των ε, αιτήσεων ασύλου φυσικά ε, βαίνει παράλληλα και με τη μεγάλη πρόκληση της ε, παροχής καταλήματος σε όλους αυτούς τους αριθμούς των μεταναστών, ιδιαίτερα στα νησιά. Έχουμε διαπιστώσει εντάσεις μεταξύ διαφορών ομάδων μεταναστών στα ελληνικά νησιά. Κομμάτι της κατάστασης είναι και αυτό. Ε, κομμάτι των προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει η ε, ευρωπαϊκή πλευρά στην Ελλάδα. Και θα ήθελα να σας δώσω κάποια στοιχεία σχετικά με τις επιχειρήσεις της Frontex. Από την 1η Ιουνίου έχουμε ξεκινήσει την επιχείρηση Ποσειδών, θαλάσσια επιχείρηση. Είχαμε την Rapid Poseidon που εξερεπνεύσε ε, το Μάιο και αντικαταστάθηκε από την τακτική Poseidon. Έχουμε υποβαθμίσει την ε, ανάπτυξη του δυναμικού γιατί ο κίνδυνος είναι μικρότερος πλέον στην Ελλάδα σε σχέση με τις ε, διελεύσεις. Βεβαίω η Frontex διατηρεί υψηλό επίπεδο ανάπτυξης δυναμικού με 550 περίπου συνοριοφύλακες δικούς μας και αυτή την εβδομάδα ε, βρίσκονται ανεπτυγμένα 19 σκάφη της Frontex στα εγχώρια δετα της Ελλάδας. Σε σχέση με την ε, κεντρική Μεσόγειο, την οδό της κεντρικής Μεσογείου, για να δώσω κάποια στοιχεία, ώστε να δείξω πώς έχουμε μετακινήσει την ε, ε, δραστηριοποίησή μας από την Ελλάδα προς τα Ιταλικά ύδατα για να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις της, στην κεντρική ε, οδό της Μεσογείου. Έχουμε περίπου 600 αεροφυλακές ε, στην Ιταλία ε, που επιχειρούν στην Ιταλία και 15 σκάφη αυτή τη στιγμή στην επιχειρησιακή ζώνη τρίτων. Αλλά πρέπει να σημειώσω ότι κάθε μέρα τα σκάφη της Frontex βγαίνουν από την επιχειρησιακή ζώνη και πλησιάζουν τα λιβικά, τις λιβικές ακτές προκειμένου να προβούν σε επιχειρήσεις διάσωσης, έρευνας και διάσωσης. Αυτά ως προς τις θαλάσσιες επιχειρήσεις και θα ήθελα ολοκληρώνοντας να αναφερθώ και στα χερσαία σύνορα. Διότι έχουμε και αυτές τις λεγόμενες ευέλικτες επιχειρήσεις αναπτύξει πλέον για να στηρίξουμε τα υποψήφια κράτη ή κράτη-μέλη σε σημεία συνόρων Βουλγαρίας-Τουρκίας, σε παραδείγματι προσερβία και έχουμε αναπτύξει τέτοιου είδου δραστηριότητες και στην Ουγγρική πλευρά στην Κροατία, στην Ελλάδα βεβαίως, με στόχο να συμβάλλουμε και στην ε, παρακολούθηση των συνόρων, στη των συνόρων, αλλά και στην υποστήριξη των ε, τακτικών ε, διελεύσεων, των τακτικών σημείων διέλευση καλύτερα. Και εκεί λοιπόν έχουμε φύλακες. Και έτσι για να ολοκληρώσω, θα ήθελα να αναφερθώ στη συνεργασία μεταξύ Frontex και χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και Τουρκίας. Έχουμε μια συμφωνία συνεργασίας συνάψη με, όλα τα δυτικά, με όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, Βοσνία, Ριζεγοβίνη, Σερβία, Μαυροβούνιο, Πρόσφατα υπέγραψα και συμφωνία συνεργασίας με το Κοσφοπέδιο. Επίσης, συμφωνία συνεργασίας έχουμε με την πρώην Δημοκρατία της Μακεδονίας και με την Αλβανία. Ε, με την Τουρκία έχουμε μνημόνιο συνεννόησης, Memorandum of Understanding, και με τις ε, χώρες αυτές στο σύνολό τους ε, προσπαθούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία. Σας δώσω ένα παράδειγμα λοιπόν σε σχέση με την Τουρκία. Όρισα, ε, διόρισα έναν ε, σύνδεσμο ε, της Frontex ε, στην Άγκυρα. Τον όρισα λοιπόν την 1η Απριλίου, είναι κατεστημένο στην Άγκυρα και η δουλειά του είναι να παρακολουθεί την, τις εργασίες των αρχών επιβολής της τάξης στην Τουρκία, αλλά και να συνομιλεί με τις ε, τουρκικές αρχές ε, εκπροσωπώντας τη Frontex για ανταλλαγή ε, πληροφοριών ή για να συμβάλλει στην, σε μια κοινή ανάλυση κινδύνου. Επίσης έχουμε εντατικοποιήσει τη συνεργασία με την νέα Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης της Μετανάστευσης που θεσπίστηκε στο τουρκικό Υπουργείο Ιστορικών πρόσφατα. Οι διευθυντές αυτή τη γενική Διευθύνσης επεσκέφθησαν την Frontex, όπως και εγώ επεσκέφθην τη Γενική Διεύθυνση το Μάρτιο στην Άγκυρα. Και προγραμματίζω μια νέα επίσκεψη τον Ιούλιο. Έχουν εντατικοποιήσει λοιπόν ε, η Frontex και οι τουρκικές αρχές την ε, συνεργασία τους και το διάλογο βέβαια. Για τις λοιπές χώρες και ιδίως ε, τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων θέλω μόνο να υπογραμμίσω ότι επί παραδείγματι σε σχέση με την Αλβανία ή τη Σερβία οργανώσαμε πρόσφατα ε, εκπαίδευση για την επαναπροώθηση έτσι ώστε και οι δύο χώρες να μπορούν τώρα πια να ξεκινήσουν να αναπτύξουν το εθνικό τους δυναμικό σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και να, οργανώνουν, ε, να μπορούν να οργανώνουν ε, ε, επιχειρήσεις επαναπρόθεσης προς τρίτες χώρες. Ολοκληρώνω λέγοντας πως η Frontex είναι κύριος παράγων στο Προενταξιακό Ταμείο ΙΠΑ, έχει αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει αναλάβει τη διαχείριση 5,5 εκατομμυρίων ευρώ που θα διατεθούν από τώρα έως το 2018 στον τομέα της ε, διαχείρισης συνόρων, ανάπτυξης δυναμικού και πολιτικές ε, επαναπροωθήσεως. Το δε προηγούμενο φθινόπορο κατά την προπαρασκευή αυτού του έργου ε, κλήθημε να το τροποποιήσουμε προκειμένου να παρακολουθήσουμε τις πρόσφατες εξελίξεις και έτσι τώρα δίνουμε περισσότερο βάρος στην ε, καταχώρηση, στο δυναμικό καταχώρηση της χώρας των Δυτικών Βαλκανίων και βέβαια στη δυνατότητα για τις χώρες αυτές να υποδεχθούν ή να αντιμετωπίσουν καλύτερα εμ, εκτεταμένες ροές μεταναστών από διαφορετικές περιοχές. Γιατί αυτό που διαπιστώθηκε πέρσι ήταν ότι οι χώρες των Νοτικών Βαλκανίων δεν ήταν χώρες προέλευσης, αλλά διέλευσης. Άρα είναι διαφορετικό τελείως το ζήτημα και πρέπει αυτές οι χώρες, χώρες Νοτικών Βαλκανίων, στη διαδικασία βέβαια προετοιμασίας για την ένταξη ως χώρες υποψήφιες, να προετοιμάζονται για την εφαρμογή των προδιαγραφών αυτών για τη διαχείριση των συνόρων. Σε ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και βέβαια είμαι στη διάθεσή σας για κάθε ερώτηση ή συζήτηση θα θέλατε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λετζέρη. Κύριε Λετζέρη. Ήταν πολύ ενδιαφέρον η παρουσίαση, πολύ ενημερωτική. Έχουμε χρόνο τώρα για ερωτήσεις, ε, παρατηρήσεις. Οπότε δίνουμε το λόγο στους προσκεκλημένους ε, για να ακούσουμε διάφορες απόψεις και να κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση. Οποιουσδήποτε από το ακρατήριο μπορεί να κάνει ερωτήσεις ελεύθερα ή παρατηρήσεις. Παρακαλώ. Έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Λεζερή. η οδός των Δυτικών Βαλκανίων έχει κλείσει σχετικά. Ποιοι παραγόντες ε, συντείνουν στο να βλέπουμε πολύ μικρούς αριθμούς ε, από την Ιβυρική οδό. Ήταν πιο ανοιχτή το 2005-2007, αλλά τώρα είναι σχετικά ήρεμα αν συγκρίνουμε με τα στοιχεία που έχουμε από την Κεντρική και την Ανατολική Μεσόγειο. Ευχαριστώ. Well, that's, uh, that's... Έχετε δίκιο. Η επωνομαζόμενη οδός των δι... της Δυτικής Μεσογείου αντιστοιχεί μόλις στο 2% του συνολικού αριθμού των παράτυπων διαλέψεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως πολύ σωστά είπατε πριν από 10 χρόνια ή 15 χρόνια είχαμε κρίση σε εκείνη την περιοχή. Ο λόγο για τον οποίο έχει σταθεροποιηθεί πλέον η κατάσταση οφείλεται σε διάφορου παράγοντε. Ένα σημαντικό παράγον είναι η σωστή συνεργασία μεταξύ Ισπανία με τρίτες χώρες και, όπως το Μαρόκο, αλλά όχι μόνο το Μαρόκο, και τις χώρες της Δυτικής Αφρικής. Υπάρχουν διαφορά κίνητρα που χρησιμοποιούνται και οικονομικά κίνητρα ώστε οι δυνητικοί μετανάστες να παραμένουν στην ε, χώρα τους. Ε, εδώ αναφέρομαι σε χώρες Δυτικής Αφρικής. Ένας άλλος παράγων είναι ότι η οδός αυτή είναι ιδιαίτερα ρεψοκινδυνευμένη από τις χώρες της Δυτικής Αφρικής μέσω του Ατλαντικού, μέσω των Κανάριων νήσων είναι μια επικίνδυνη οδός ε, και πολύ μεγάλη. Και λόγω της κατάστασης στη Λιβύη φυσικά ένα τμήμα της παράτυπης μετανάστευσης ε, κινείται τώρα από τις χώρες της Δυτικής Αφρικής προς τη Λιβύη. όπου ελπίζουν ότι θα έχουν τη δυνατότητα να περάσουν προς την Ιταλία. Δύο είναι οι εξηγήσει. Σωστή λοιπόν συνεργασία μεταξύ Ισπανίας, Μαρόκου και χωρών της Δυτικής Αφρικής. Η επικινδυνότητα και το μήκος της οδού αυτής με, μέσω της Ισπανίας αλλά και το γεγονός ότι η οδός της κεντρικής Μεσογείου φαίνεται πιο ελκυστική και εκεί φυσικά δρούν και εγκληματικά δίκτυα. Αλλά επίσης ε, τα μέσα χερσαίας μεταφοράς μεταξύ των χωρών της Δυτικής Αφρικής ε, ε, δεν είναι τόσο ακρίβεια. Αυτό βοηθά τους μετανάστες να κινηθούν μόνοι τους χωρίς να εμπλακούν με εγκληματικά δίκτυα. Άλλες ερωτήσεις? Σας ευχαριστώ με βουλευτές του Σοδημοκρατικού Κόμματος. Ε, έγινε λόγος στην προηγούμενη ομιλία για ε, απόφαση Ελλήνων δικαστών ότι δεν είναι ασφαλής χώρα η Τουρκία και άρα δεν μπορεί να γίνεται επαναπροώθηση μεταναστών εκεί. Τώρα γιατί είδους ε, ασφάλεια μιλάνε δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Ε, πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει στην Τουρκία αγώνας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Πολύ μεγάλος αγώνας. Με συγκεκριμένα και αυτά αποτελέσματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει οδήποτε ζήτημα ασφάλειας για τους μετανάστες ή τους πρόσφυγες. Η χώρα μας θεωρείται χώρα διελεύσεως. Η Ελλάδα επειδή είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε, θα πρέπει να εξετάζει τις αιτήσει ασύλου και να ε, διοχετεύει τους ε, πρόσφυγες στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αφού είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν, είπατε ότι έχετε συμφωνία και συνεργασία με τις υποψήφιες χώρες. Εγώ νομίζω ότι αποφάσεις αυτές των ε, Ελλήνων δικαστών, οι οποίες δείχνουν προκατάληψης βαρούς Τουρκίας, ε, μπορείτε να μας εξηγήσετε αν έδωσαν μια, ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ε, κύριε Λεζερή, μπορείτε να απαντήσετε. Well, uh... Maybe next few questions and... Να ακούσουμε ίσως λίγες ακόμη ερωτήσεις. Παρακαλώ. thank you. My name is assistant of... Ευχαριστώ. Είμαι βοηθός του κύριου Κενά. Ερώτηση προς τον κύριο Λεζερή. Ευχαριστούμε για την ενδιαφέρουσα ομιλία σας. Το έργο της Frontex είναι πολύ σημαντικό η ερώτησή μου είναι η εξή. Είναι πολύ σημαντικό να βοηθάμε τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και από την άλλη να μειώσουμε την τεράστια ροή οικονομικών μεταναστών. Επίσης είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τη διάσωση στη θάλασσα. Πρέπει να προσφέρουμε ρογή σε πλοία και ανθρώπους που κινδυνεύουν στη θάλασσα. Αλλά η ερώτησή μου είναι η εξή. Αυτή τη στιγμή μήπως η Frontex άθελά προωθεί κατά κάποιο τρόπο την εισρωή ε, παράτυπων μεταναστών, διασώζοντας ανθρώπους ε, στη Μεσόγειο χωρίς να τους επιστρέφει στην ε, Λιβύη ή την Αίγυπτο, αλλά φέρνοντας στην Ιταλία. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το όνομά μου είναι από το Αφιόν Καραχισάρ. Κόμμα Τουρκία. Ε, είπατε ότι έχει υποδεχθεί 2 εκατομμύρια πρόσφυγες στην Τουρκία. Δεν είναι σωστό, είναι 3 εκατομμύρια και πάνω. 2,7 από τη Συρία και μετά επιπλέον από το Ιράκ, το Αφγανιστάν κτλ. Ο αριθμός των προσφύγων συνολικά στην Τουρκία ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια και είναι δεκαπλάσιος του συνόλου των προσφύγων που έχουν υποδεχθεί χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάντως για τις αντικειμενικές διαπιστώσεις οποίες εκφράσατε μέσα από την ομιλία σας. Ε, η συμβολή της Τουρκίας στην υπόθεση αυτή και ιδιαίτερα μετά τη Συμφωνία Επανεισδοχής νομίζω ότι έχει βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση, σχεδόν εκμηδενισμό των μεταναστευτικών ροών προς την Τουρκία. Είναι τεράστια η προσπάθεια που έχει καταβάλει η Τουρκία προς την κατεύθυνση αυτή και εμείς έχουμε δαπανίσει πάνω από 10 δισεκατομμύρια ε, ευρώ ε, δολάρια στην ε, προσπάθεια αυτή και συνεχίζουμε να δαπανούμε πολύ ψηλά ποσά και βέβαια πιστεύω ότι θα πρέπει να επικροτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ηθικά αλλά και υλικά βεβαίως στην προσπάθεια αυτή της Τουρκίας. Γιατί ε, ενώ δεν έχουμε αφήσει να φύγουν προς τα ευρωπαϊκά κράτη αυτοί οι πρόσφυγες ε, και τους έχουμε κρατήσει στη χώρα μας όπου τους υποδεχόμαστε και δαπανούμε τόσα χρήματα για να τους φροντίσουμε, έχουμε ακόμα και από την εσωτερική αντιπολίτευση ε, επικρίσεις ότι δεν ε, κάνουμε αυτό που οφείλαμε. Νομίζω όμως ότι είναι ξεκάθαρη η κατάσταση και για να περάσω σε ένα άλλο θέμα πρέπει να τεθεί ένα τέρμα σε αυτόν τον άδικο πόλεμο για να σταματήσουν να φεύγουν από τις πατρίδες τους οι πρόσφυγες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, προσπαθεί να πει στα τουρκικά ο πρόεδρος, αλλά δεν τα πολύ καταφέρνει. Θα μιλήσω από εδώ και μπρος στις, ε, στα αγγλικά. Παρακαλώ να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά την ε, εφαρμογή της, ε, της ε, Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας από αριθμητικής απόψεως υπάρχουν δύο είδη αριθμών που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Τον αριθμό των μεταναστών που δεν έχουν φύγει από την Τουρκία γιατί Υπάρχουν περισσότερες ε, περιπολίες τώρα στα τουρκικά ύδατα, αλλά και γιατί ε, υπάρχουν περισσότερες περιπολίες και στην ενδοχώρα στην Τουρκία. Μπορούμε απλώς να συγκρίνουμε τις ροές που είχαμε κατά τους τελευταίους μήνες και την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που είναι περίπου μηδέν, γιατί 50 αφήξει ημερησίω σε, μια σε σύγκριση με κατάσταση κατά την οποία είχαμε περίπου 2.000, 5.000, 8.000 σε κάποια στιγμή ημερησίω, είναι τεράστια διαφορά. Πρόκειται λοιπόν για μια κατάσταση που έχει μειωθεί στο μηδέν ε, σχεδόν. Από τη μία λοιπόν υπάρχει εφαρμογή της ε, δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και αυτό είναι ο ένας τρόπος να προσμετρήσει κανείς ε, την προσπάθεια που έχουν κάνει οι τουρκικές αρχές προκειμένου να ε, διαχειριστούν καλύτερα ε, το δυτικό εξωτερικό σύνορό τους, αλλά επίσης και να αποφευχθεί ότι οι μετανάστες διακινδυνεύουν τη ζωή τους. Ένα ακόμη αριθμητικό στοιχείο είναι ο αριθμός ε, των ε, μεταναστών ε, που η Τουρκία, που η, Ελλάδα θα μπορούσε να επιστρέψει στην Τουρκία. Υπάρχει όμως μία συμφόρηση εκεί πέρα στη διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα και γι' αυτό το λόγο έχουν επιστρέψει λιγότερο από 500 μετανάστες στην Τουρκία. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι επιβραδύνεται ε, και γι' αυτό το λόγο ένα άλλο τμήμα της δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας το «ένας για έναν». Ένας ε, σύρος ε, μπορεί να μετεγκατασταθεί από την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε φορά που ένας μετανάστης επιστρέφει από την Ελλάδα στην Τουρκία. Υπάρχει όμως και μια ποσοτική αύξηση, η οποία, μια ποιοτική αύξηση, η οποία δεν μπορεί να προσμετρηθεί ποσοτικά, που είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, κάτι το οποίο είχε πολύ θετικό αντίκτυπο στην καταπολέμηση των εγκληματικών δικτύων και των απειλών ε, κατά της ασφάλειας. Όσον αφορά τώρα το ερώτημα που αφορά τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων ε, περιπολίας της Frontex στην Κεντρική Μεσόγειο, αυτό το ζήτημα ε, έχει συζητηθεί πολλές φορές και νομίζω ότι η Ιταλία όταν, ε, όταν υπήρχε αυτή η επιχείρηση Mare Nostrum. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Frontex μέχρι τώρα έχουν καταφέρει να ε, βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ των ε, τριών ε, συγκρουόμενων υποχρεώσεων. Πρώτον, δεν μπορούμε να αφήνουμε τον κόσμο να πεθαίνει στη θάλασσα. Υπάρχει λοιπόν ένα ανθρωπιστικό, μια ανθρωπιστική υποχρέωση, αλλά επίσης συνάδει και με το δίκαιο της θάλασσας και με ε, το διεθνές δίκαιο. Κάθε φορά που υπάρχουν άνθρωποι σε δύσκολη κατάσταση στη θάλασσα, πρέπει να τους αναζητήσουμε και να τους διασώσουμε. Από την άλλη, πρέπει να καταστεί σαφέ ότι δεν θέλουμε να ενθαρρύνουμε εγκληματική δραστηριότητα. Αυτό είναι κάτι που δεν είναι καινούριο είναι κάτι που έχει υποθεί πολλές φορές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ ως εκτελεστικός διευθυντής της Frontex είχα κατά τον τελευταίο μήνα και κατά τον τελευταίο χρόνο το τονίσω αυτό, ότι δεν πρέπει να ενθαρρύνουμε το έγκλημα και πρέπει να αποφύγουμε οι εγκληματικές οργανώσεις να οργανώνουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο ε, βάσει της βεβαιότητας ότι θα περάσουν ε, ε, οι μετανάστες από τη Λιβύη στην Ιταλία. Υπάρχουν λοιπόν συγκρουόμενες ε, υποχρεώσεις και καθήκοντα. Αλλά τώρα για ποιο λόγο δεν μπορούμε να τους εκφορτώσουμε να τους αποβιβάσουμε στην Λιβύη είναι λόγω της αρχής της μη επαναπροώθησης. Ενδεχομένως να έχετε διαβάσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, Compact περιεκτική συνεργασία με τρίτες χώρες ε, ώστε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με οικονομική ανάπτυξη, ανάπτυξη του κράτους δικαίου, δικαίου στις χώρες προέλευσης και στις χώρες ε, διέλευσης. Δεν δίνεται όμως ε, η δυνατότητα συνεργασίας για την κατάσταση στη Λιβύη όπως ε, υπάρχει μεταξύ Μαρόκου και Ισπανίας. Απέχουμε πάρα πολύ από αυτό. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λεζερή για τις απαντήσεις σε αυτό και σε άλλα ερώτηματα και ευχαριστούμε και για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Θα ήθελα τώρα να καλέσω την κυρία Μαρίκα στην Βέρζια μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισηγήτρια για θέματα μετανάστευσης και ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Υποεπιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Παρεπιπτόντως, η κυρία Βερζιά είναι ε, μία από τα, ένα από τα πιο δραστήρια μέλη επί του ζητήματος. Ε, κύριε Βεζιά, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που σας έχουμε εδώ. Έχετε τον λόγο. Merci. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν έχω τη μεγαλύτερη επιρροή αλλά σίγουρα εδώ και πάρα πολύ καιρό με ενδιαφέρουν τα ζητήματα αυτά. Είμαι μέλος της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ταυτόχρονα μέλος ε, της Επιτροπής ε, Πολιτικών Ελευθεριών. Η εμπειρία μου δηλαδή εντός του Κοινοβουλίου αφορά εργασία ε, εσωτερικής αλλά και εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο ώστε να επιτύχουμε, όπως το λέμε πολύ συχνά εδώ, μια ολιστική προσέγγιση των μεταναστευτικών πολιτικών. Χθε ήταν η Παγκόσμια Μέρα των Προσφύγων και η UNHCR δημοσίευσε μια νέα έκθεση. Όταν λέμε λοιπόν ότι είναι άνευ προηγουμένου η μεταναστευτική κρίση, η προσφυγική κρίση, θέλω να αναλύσω λίγο την κατάσταση. 65 εκατομμύρια εκριζωμένοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι. Αυτό σημαίνει μετατοπισμένοι και πρόσφυγες. Ε, το 85% αυτών των ανθρώπων βρίσκονται σε ε, αναπτυσσόμενες χώρες. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ήπειρο στο σύνολό της, δεν στέκεται στο ύψος ε, των περιστάσεων αυτής της παγκόσμιας κρίσης που πλήττει τον πλανήτη. Για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ήπειρος ε, δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, διότι αντί να προσπαθεί να απαντήσει, να δώσει μια λύση σε αυτή την κρίση, κλείνουμε όλο και περισσότερο τα σύνορά μας. Περιφρονώντας ε, το διεθνές δίκαιο και τις Διεθνές συμφωνίες, όπως υπενθυμίζεται από το UNHCR, και από τα Ηνωμένα Έθνη. Ε, αναφέρομαι σε ανθρώπους βέβαια οι οποίοι ασχολούνται όπως εδώ σε αυτή την αίθουσα με την πολιτική γειτονία και θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν οι υποχρεώσεις που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από εσάς επί του θέματος περιλαμβάνουν την τήρηση των διεθνών συμφωνιών, την υπογραφή διεθνών συμφωνιών και κυρίως εκείνων ε, που αφορούν το ζήτημα αυτό, τη συνθήκη της Γενέβης, τη Διεθνή Συνθήκη Δικαιωμάτων του Παιδιού, τη Διεθνή Συνθήκη για τα Δικαιώματα των Γυναικών, μεταξύ άλλων. Δεν αρνούμε τις προσπάθειες της Frontex, παρότι πολλοί επικρίνουν τη Frontex. Εγώ όχι θεωρώ ότι το βασικότερο πρόβλημα που έχουμε είναι η απουσία ευρωπαϊκού οράματος όσον αφορά αυτά τα ζητήματα. Κάθε κράτος μέλος βλέπει την μεταναστευτική πολιτική από τη δική του οπτική γωνία. Ενώ στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα ε, τα πράγματα διαφέρουν από χώρο σε χώρα. Οι πληθυσμοί που φτάνουν ε, σε κάθε χώρα είναι διαφορετικοί. Οι ιστορίες των μεν και των δε μπορεί να διαφέρουν σημαντικά. Εγώ είμαι Γαλλίδα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα από τη χώρα μου. Η Γαλλία είναι η χώρα που έχει την παλαιότερη μεταναστευτική ιστορία στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Γιατί την παλαιότερη, διότι ξεχνάμε συχνά ότι από το 1850 και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια Ευρωπαίων ε, μετανάστευσαν σε ολόκληρο τον κόσμο και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Η Γαλλία έχει μια ιδιαίτερη ιστορία διότι είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που άλλαξε τη μεταναστευτική ισορροπία, δηλαδή όπου οι μετανάστες που εισέρχονταν στη χώρα έγιναν ξαφνικά περισσότεροι από αυτούς που έβγαιναν από τη χώρα. Και οι γειτονικέ χώρες, Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία, αλλά και οι Πολωνοί και οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι μετανάστευσαν. Μετά μόνο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έκανε έκκληση η Γαλλία στις απικίες της για να επανοικοδομήσει την Γαλλία. Η Γαλλία μου λοιπόν χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από αυτά τα ιστορικά στοιχεία. Η πρώτη ε, ξένη κοινότητα σε γαλλικό έδαφος ήταν η Πορτογαλική πριν από κάθε άλλη. Και κάθε χώρα χαρακτηρίζεται από αυτό και η Μεγάλη Βρετανία έχει μια ιστορία με την κοινοπολιτεία. Όταν ακούμε τις συζητήσεις για το Brexit σήμερα και την καταπολέμηση της μετανάστευσης, αυτή δεν στρέφεται κατά των ε, υπηκών ε, της κοινοπολιτείας, αλλά κατά της Ανατολικής Ευρώπης. Κάθε χώρα λοιπόν έχει την ιστορία της και εμείς ως Ευρωπαίοι έχουμε μια ευθύνη να οικοδομήσουμε μια κοινή ιστορία, να χρησιμοποιήσουμε από κοινού τα καλύτερα στοιχεία που έχουμε. Ενώ εδώ βλέπουμε να γίνεται ακριβώ το αντίθετο τα κράτη-μέλη μας, επειδή η ευθύνη, όπως είπατε πολύ σωστά, στο πλαίσιο της Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, είναι ευθύνη του Συμβουλίου των Κρατών Μελών. Και εδώ μιλάμε για δήλωση και όχι συμφωνία, διότι αν είχε υπάρξει διεθνή συμφωνία, πραγματικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει γίνει προσφυγή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, γεγονός που δεν συνέβη. Να αναφέρω και κάτι άλλο, συγκριτικά, εσείς προέρχεστε από πολλές χώρες που ζητάτε ε, συμφωνίες ε, απελευθέρωσης των θεωρήσεων. Και εγώ είμαι σκιώδη εισηγήτρια για το θέμα αυτό στη δική μου ομάδα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για μένα πρέπει να υπάρχει μια συνοχή μεταξύ όλων αυτών. Όταν γίνεται αίτηση ε, προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή για απελευθέρωση των θεωρήσεων ε, ε, και εκεί πρέπει να τηρούνται τα ίδια κριτήρια και μόνο με συνεργασία μεταξύ μας μπορούμε να προχωρήσουμε. Ενώ τι συμβαίνει τώρα όσον αφορά τη Συμφωνία Απελευθέρωση των Θεωρήσεων, λαμβάνουμε απαντήσει καθαρά πολιτικέ. Ορισμένοι λένε ναι, ορισμένοι λένε όχι. σε άλλα θέματα και κανεί δεν καταλαβαίνει γιατί. Οπότε και εκεί πρέπει να προχωρήσουμε λίγο με πιο ανοιχτά χαρτιά. Το άλλο στοιχείο είναι ότι πιστεύω πως σφάλουμε όταν προσπαθούμε να διαχωρίσουμε τους καλούς πρόσφυγες και τους λοιπούς μετανάστες. Ναι, δεν είναι όλοι οι οικονομικοί μετανάστε και μπορούμε να επανέλθουμε στο ζήτημα των οικονομικών μεταναστών, αλλά αυτό που κάνουμε, ειδικότερα στο πλαίσιο του ένα προ ένα με την Τουρκία, προσπαθούμε να έχουμε μια συμφωνία όπου διαχωρίζουμε του καλού πρόσφυγε, αυτού που έρχονται από τη Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν, διότι τους αναγνωρίζεται ένα δικαίωμα ασύλου σε ευρωπαϊκές χώρες περισσότερο και τους λοιπούς. Δεν είναι τρόπος αυτός ε, τήρησης του διεθνούς δικαίου, σωστός. Και το κάθε κράτος μέλος έχει άλλες πρακτικές. Αυτό που εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι τόσο για τις πρόσφυγες σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και για τους ανθρώπους που ε, περνούν τη Μεσόγειο, έχουμε όλο και περισσότερες γυναίκες, όλο και περισσότερα παιδιά. Σε παγκόσμιο επίπεδο, από τα 65 ε, εκατομμύρια προσφύγων, η μισή είναι παιδιά. Από αυτούς που περνούν τη Μεσόγειο, το 1 τρίτο είναι παιδιά. 1 τρίτο είναι γυναίκες. Ενώ πριν από μερικά χρόνια ήταν το αντίστροφο. Ήταν 60% άντρες τότε. Σήμερα έχουμε 60% γυναίκες και παιδιά. Και παιδιά όλο και πιο μικρά παιδιά όλο και περισσότερο ασυνόδευτα. Εγώ πήγα στην Ιταλία πριν από μερικές εβδομάδες στο ε, κέντρο του Ποτσέλο και οι υπεύθυνοι του κέντρου μου είπαν ότι είχαν ε, συγκλονιστεί από την άφηξη μόνων παιδιών. Ένα κοριτσάκι 9 χρονών είχε περάσει τη Μεσόγειο μόνο του, μου είπαν. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί για το Compact που θα θέλαμε να γίνει μια σωστή αξιολόγηση της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας πριν ε, αρχίσουμε να διαπραγματευόμαστε με τις χώρες καταγωγής. Ξέρετε, οι χώρες καταγωγής και αυτές έχουν να αντιμετωπίσουν τρομακτικές καταστάσεις όσον αφορά τη μετανάστευση. Και όπως πολύ σωστά είπατε, έχουμε και μια ανθρωπιστική υποχρέωση σε θέματα διάσωσης στη θάλασσα. Και εγώ διαπιστώνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε 5 εκατομμύρια για τη διάσωση στη θάλασσα. Αναφερθήκατε στο Μαρενόστρουμ. Το Μαρενόστρουμ ε, είχε προπολογισμό 95 εκατομμύρια μόνο από την Ιταλία. Υπάρχουν θέματα λοιπόν ευθύνης διαφορετικά. Όσον αφορά τη διάσωση στη θάλασσα, το 1 τρίτο γίνεται από την εμπορική ναυτιλία. Το 1 τρίτο των διασώσεων. το εμπορικό ναυτικό. Για να μην μιλήσουμε για τις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις που διασώζουν χιλιάδες και χιλιάδες ανθρώπων. Δεν λέω ότι η ακτοφυλακή δεν σώζει κόσμο, σίγουρα, αλλά ξέρετε ο αριθμός θανάτων των νεκρών συνεχίζει να αυξάνεται. Είμαστε ε, στη Μεσόγειο, έχουμε ξεπεράσει τις 30.000 την τελευταία 15, ετία. 1.370 είχαμε στη Μεσόγειο, γυναίκες, παιδιά. 3.170 πέρυσι, πάνω από 2.500 σήμερα, μέχρι σήμερα φέτος. Ε, συγγνώμη που αναφέρομαι σε ρεκόρ, αριθμό σε αριθμό ρεκόρ πέρυσι, μέχρι τα τέλη του χρόνου θα έχουμε ξεπεράσει τις 7.000 στη Μεσόγειο και όπως αναφέρατε ακολουθούν οδούς όλο και πιο επικίνδυνες. Φεύγουν όλο και πιο συχνά από την Αίγυπτο προς την Ιταλία, δηλαδή ταξίδι 13 ημερών για να, διέλθουν, για να περάσουν τη Μεσόγειο ή περνούν από τη Λιβύη όπου πέφτουν θύματα της εμπορίας ανθρώπων διότι δεν υπάρχει πλέον κράτος δικαίου στη Λιβύη. Όσο περισσότερο εμείς κλείνουμε τα σύνορα τόσο περισσότερο τροφοδοτούμε την παράνομη διακίνηση. Όσα αστυνομικά μέτρα και να λάβουμε οι διακινητές και οι έμποροι θα βρίσκουν πάντα άλλες οδούς και θα θέτουν τη ζωή αυτών των ανθρώπων όλο και περισσότερο σε δίκαιο. Αυτό είναι ανεύθυνο και ανάξιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να τελειώσω, ε, είπατε πολύ σωστά κύριε Πρόεδρε, ναι, πρέπει να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δει τη δημογραφική και την οικονομική της κατάσταση. Δημογραφικά η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μετανάστες. Οι περισσότερες χώρες αυτές σήμερα οφείλουν τη δημογραφική τους ανάπτυξη μόνο στην παρουσία των μεταναστών. Η Γερμανία θα έλεγα σχεδόν ε, ότι είναι μοντέλο παρότι δεν συμφωνώ απόλυτα, δεν έχω ως πρότυπο την κυρία Μέρκελ, αλλά η Γερμανία βρίσκεται σε δημογραφική και οικονομική θέση που είναι η πιο χαρακτηριστική. Η ηλικιακή πυραμίδα είναι εντελώς αντίστροφη σε σχέση με σχέση με τις πραγματικές δημογραφικές ανάγκες. Και αυτό εξηγεί εν μέρη τη στάση της Γερμανίας πέρυσι γιατί η κυρία Μέρκελ είναι Γερμανίδα από την Ανατολική Γερμανία και είναι και κόρη ιερέα. Και όλα αυτά δημιουργούν μια νοοτροπία, μια ηθική πολύ διαφορετική. Για ποιο λόγο να αντιδρούσε διαφορετικά η Γερμανία διότι στο παρελθόν όσον αφορά την υποδοχή των προσφύγων οι συνθήκε στη Γερμανία ήταν φρικτέ. Πάντα σκεφτόμαστε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ξεχνάμε τι έγινε μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου 12 εκατομμύρια Γερμανοί επανήλθαν στη Γερμανία και έτσι όπω είχαν τα πράγματα στη Γερμανία τότε, αυτό σημάδεψε την ιστορία τη Γερμανία. Οπότε σα λέω, κάθε χώρα αντιδρά βάσει τη δική τη ιστορία. Μου κάνει εντύπωση όταν ακούω δηλώσει από χώρε ε, που ε, που βρίσκονται πολύ κοντά στην Τουρκία, οι οποίε βρίσκονται υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι ιστορίε του είναι πολύ διαφορετικέ γιατί η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν ε, είχε την ίδια πολιτική με τι διάφορε χώρε. Όλα παίζουν ρόλο στην οτροπία και πιστεύω την ευθύνη ενό πολιτικού να μιλήσει διαφορετικά να μην επιτρέπει να ανεβαίνει ο φόβο, αλλά να κάνει μια υπεύθυνη συζήτηση σε σχέση με τι δημογραφικέ και οικονομικέ ανάγκε. Και θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται του ε, μετανάστε. Όχι να ανοίξει διάπλατα τα σύνορα, απλά να έχει μια πολιτική υπεύθυνη επί του θέματο και να ανοίξει νόμιμες οδούς μετανάστευσης όπως το ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως το ζητά η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου εδώ, του Ευρωκοινοβουλίου, να μην κάνουμε διαχωρισμό των καλών προσφύγων από τους κακούς οικονομικούς μετανάστες δεν είναι σωστό, δεν είναι ρεαλιστικό όσον αφορά το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ήπειρος γυράσκουν σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο και ευθύνη μας ως πολιτικών είναι να είμαστε ανοιχτό ανοιχτόμυαλοι ως προς τον κόσμο αντί να κλεινόμαστε στον εαυτό μας. Στην Ευρώπη έχουμε μια τεράστια ιστορία, μια όμορφη ιστορία Εμένα ε, μου αρέσει πάρα πολύ η ευρωπαϊκή ιστορία. Βλέπω τις καλές πλευρές αλλά και τις κακές και πιστεύω ότι πρέπει να την αξιοποιήσουμε ώστε οι συζητήσεις που κάνουμε να συμμορφώνονται με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Και τώρα Ας ακούσουμε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Από το, από το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου και μέλος της Επιτροπής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Ελευθεριών. Ένα σύντομο σχόλιο. Στα όσα είπε η κυρία Βερζιά. Πιστεύω ότι η ομιλία αυτή είναι η καλύτερη από αυτές που άκουσα αυτό το διήμερο. Πολύ ρεαλιστική, σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Εμείς στο Μαυροβούνιο την Ευρώπη τη βλέπουμε πάνω απ' όλα σαν μια Ευρώπη των αξιών. Προσπαθούμε τις αξίες μας, τι ευρωπαϊ... τις βαλκανικές αξίες, να τις αλλάξουμε και να δείξουμε προστερή αλληλεγγύη, ευθύνη, υπευθυνότητα, ανθρώπινα δικαιώματα που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή στο βαθμό αυτό στη χώρα μας. Η ομιλία σας ήταν συναρπαστική και πολύ ρεαλιστική. Πάνω απ' λοιπόν. Πρέπει να ξεκινήσω λέγοντα ότι δεν έχει τόσο σοβαρά προβλήματα με τη μετανάστευση στο Μαυροβούνιο. Αυτό είναι το ένα. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο κοινωνικό ή οικονομικό. Είναι χαρακτηριστικά πολιτικό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαρακτηριστικά πολιτικό. Εάν λοιπόν θέλουμε να μιλήσουμε ξεκάθαρα για τις ε, αιτίες και τις συνέπειες, η αιτία είναι ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια, αλλά πολλά χρόνια πριν. Ο πόλεμος στο Ιράκ το 2003, του Αφγανιστάν το 2001 της Συρίας πριν από τρία χρόνια. Όλοι αυτοί οι πόλεμοι, όλα αυτά τα προβλήματα οφείλονται στο ότι, έτσι πιστεύω εγώ προσωπικά, το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι δεν έχει εξωτερική πολιτική με ε, διάσταση άμυνας. Πρέπει να έχει πολύ πιο δραστήρια ε, εξωτερική πολιτική η Ευρωπαϊκή Ένωση και να προσπαθήσει να να προσπαθεί να δίνει λύσεις σε διάφορε περιοχέ, γιατί είναι πολλέ αυτέ οι οποίε εκδηλώνονται προβλήματα και στη Βόρεια Αφρική, συνεπιφέροντας και εσωτερικέ αλλαγέ στι χώρε. Εάν ε, μείνει να παρακολουθεί την κατάσταση μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση και να περιμένει να φτάσουν τα προβλήματα στα σύνορά τη, δεν νομίζω ότι θα έχει κάνει ευφύ επιλογή. αυτά τα οποία συμβαίνουν στις ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι συμβατά με τις ευρωπαϊκές αξίες. Εδώ θα σταματήσω το σχολείο μου, εκφράζοντας πλήρη υποστήριξη στα όσα είπατε. και ελπίζοντας ότι μαζί με τους λοιπούς βουλευτές θα βρείτε κοινό πεδίο συνεννόησης και ιδέες για την προαγωγή των πραγματικών ευρωπαϊκών ιδεουδών, όχι μόνο επί χάρτου ή μέσα από τις δηλώσεις, αλλά κατά τρόπο απτό. Σας ευχαριστώ θερμά. Φαλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λιζόλη, σχόλια. Ναι, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θέλω απλώ να ενημερώσω τα στοιχεία τα σχετικά με τις θαλάσσιες επιχειρήσεις της Frontex μετά την περσινή τραγωδία, την τραγωδία του Απριλίου του 2015, με 800 περίπου νεκρούς στην Κεντρική Μεσόγειο μέσα σε ένα, με ένα ναυάγιο μόνο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να τριπλασιάσει τον προπολογισμό των θαλασσίων επιχειρήσεων της Frontex και έτσι για το 2015 ο προϋπολογισμός για θαλάσσιες επιχειρήσεις ήταν 67 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο 2015. Για φέτος 102 εκατομμύρια ευρώ προβλέπονται ειδικά για τις θαλάσσιες επιχειρήσεις της Frontex, συγκεκριμένη δηλαδή υποστήριξη των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Από την 1η Ιανουαρίου φέτος έχουμε προβεί σε έρευνα διάσωση 50.000 μεταναστών. 35 στο Αιγαίο, 35.000 στο Αιγαίο μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας και 15.000 μέχρι τώρα στην Κεντρική Μεσόγειο. Αυτά για να σας δώσω τα τελευταία στοιχεία τα σχετικά με τον προϋπολογισμό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ιδιαίτερα θα ήθελα να αναφερθώ στις ε, προτάσεις του νομιλητών μας σε σχέση με την περιγραφή του προβλήματος και, το, και των συμπερασμάτων ε, και τις προτάσεις λύσεων ε, που ακούσαμε. Ιδιαίτερα έγινε λόγος για αδυναμία εξέβρεσης λύσης. Νομίζω ότι θα πρέπει ίσως να κοιτάξει για την κάθε χώρα ε, η κάθε χώρα μάλλον, τι είδους συνθήκες επικρατούν και συγκυριακά ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις εξελίξεις, αντί να προσπαθούμε να επιβάλλουμε μόνο κόμματα μία λύση. Και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική η αναγνώριση πολλαπλών διαστάσεων στο πρόβλημα. Η Τουρκία βεβαίως έχει συμμετάσχει σε πολλές ε, συνόδους κορυφή στις 18 Μαρτίου του 2016 ε, την τελευταία, όπου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης έγινε ανάλυση και διαπίστωση της κατάστασης Η Τουρκία βεβαίως παραμένει πάντοτε πιστή σε όλες τις δεσμεύσεις της, διεθνείς ε, συμφωνίες και συμβάσεις και τις ε, Η φόρμουλα ένας προς έναν για τους ε, πρόσφυγες, ε, μετανάστες, ε, ξεκινάει με την ε, πρόταση ένας ε, Σύρους μετανάστης να γίνεται δεκτός στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένας να επιστρέφεται. Βεβαίως πάντοτε ξεκινάμε με τα προγράμματα της, του εθελοντικού επαναπατρισμού. Ε, υπάρχει η επιδίωξη πάντοτε εξασφάλισης συνθήκων ομαλής διαβίωσης για τους Σύρους μέσα στα σύνορα της Συρίας. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το τονίσουμε ιδιαίτερος και να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση ώστε να συμβάλλουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Από τις διαπιστώσεις που ακούστηκαν επίσης ήταν το θέμα της ε, ανάγκης για ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για την ε, κατάρριξη της υποχρέωσης θεώρησης διαβατηρίων για Τούρκους υπηκός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για μας, είναι κοινά τα κριτήρια και η μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί και βεβαίως θα υπαχθούμε σε αυτά και θα εκπληρώσουμε τους ε, όρους θεωρούμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευρά τη πρέπει να προχωρήσει σε συγκεκριμένα βήματα σε ο βαθμό που τους αντιστοιχούν οι υποχρεώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Uh, thank you and uh, our from uh, Greece, from Ευχαριστώ πολύ συνάδελφος από την Ελλάδα. Εύη Καρακώστα, βουλευτής της, ε, του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ε, ήθελα πραγματικά να συγχαρώ την κυρία Βερσά για την εισήγησή της. Ήταν πραγματικά εξαιρετική. Όπως και αρκετές χθεσινές ε, εισηγήσεις ήταν στο ίδιο πλαίσιο. είναι αλήθεια ότι μπαίνει το μεγάλο ερωτηματικό αν θέλουμε ανοιχτά σύνορα ή κλειστά σύνορα και σε ποιο βαθμό ελέγχουμε αυτά. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι στην Ελλάδα, παραδείγματο χάρη, έχουν, έχουν, από την Ελλάδα έχουν επιστραφεί 462 πρόσφυγες προς την Τουρκία, οι οποίοι απλά δεν ζήτησαν άσυλο. Είναι αυτοί δηλαδή ε, οι άνθρωποι που θέλησαν να γυρίσουν προς την Τουρκία. Είναι πολύ μικρός όμως ο αριθμός αυτός και πραγματικά πολύ σωστά θέσατε κύριε Λετζέρη το ερωτηματικό γιατί τόσος μικρός αριθμός ε, ζητά <clears throat> αυτή την επαναεισδοχή. Εκείνο βεβαίω που πρέπει να εξετάσουμε επίση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποσχεθεί ότι θα έπαιρνε 6.000 πρόσφυγε το μήνα. Σε, ε, γενικά και τον προηγούμενο πήρε, μήνα πήρε μόνο 780, αν θυμάμαι καλά. Ε, αυτά είναι νούμερα τα οποία πρέπει να τα ελέγξουμε. Πραγματικά πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα και των επιπλέον προσφύγων που μένουν στην Ελλάδα. Ε, είναι, ε, ίσως θα πρέπει να βρεθούν και νέε νέες συμφωνίες αν πραγματικά μπορούν να φεύγουν πρόσφυγες κατευθείαν από την Ελλάδα όπως είναι η επανένταξη οικογενειών, ε, να ελέγξουμε τα συνόδευτα παιδιά και προς ποια κατεύθυνση πηγαίνουν και πώς τα προφυλάσσουμε από το διεθνές εμπόριο. Πάντως, πραγματικά, στην κατεύθυνση που έβαλε η κυρία Βερσά, πρέπει να ελέγξουμε το πόσο πραγματικά ενδιαφερόμαστε για τους ανθρώπους ε, και όσο διαρκούν οι πόλεμοι που εμείς θα θέλαμε να φροντίσει το σύνολο της Ευρώπης να σταματήσουν οι πόλεμοι στις χώρες τους, να, να σταματήσουν οι κακές οικονομικές συνθήκες στις χώρες τους, γιατί νομίζω ότι κανείς δεν θέλει να φύγει από την πατρίδα του χωρίς να έχει προβλήματα. Ε, έτσι και από την Ελλάδα έχουν φύγει μετανάστες, δηλαδή ο ελληνικός πληθυσμός ανά τον κόσμο είναι διπλάσιος από αυτόν που έχουμε στη χώρα μας. Ε, και πολύ σωστά ετέθη, αλλά ε, ανάγκες ε, βρίσκονται, όπως τώρα φεύγουν από την Ελλάδα εξαιρετικοί επιστήμονες. Έχουμε δηλαδή εξαγωγή επιστημόνων και συγχρόνως έχουμε ένα μεγάλο αριθμό προσφύγων. Είναι η ανταλλαγή πληθυσμών είναι σοβαρό θέμα, πρέπει να είναι ανοιχτό κατά τη γνώμη μας ε, και βέβαια κυρίαρχο στη σκέψη μας είναι το πώς χωρίς να κλείνουμε σύνορα ε, να γίνεται αυτή η διακίνηση με κανόνες για να μην έχουμε νεκρούς πραγματικά στη θάλασσα γιατί πολύ καλά κύριε Λετζέρη είπατε ότι κλείνοντας ε, το Αιγαίο, τα σύνορα, τα σύνορα δηλαδή των Σκοπίων με την Ελλάδα κλπ αναγκάζουμε τους διακινητές να πηγαίνουν προς πολύ πιο δύσκολους διόδους προς πολύ πιο δύσκολα περάσματα για την ανθρώπινη ζωή. Αυτό ήθελα να δούμε και αν μπορέσουμε να βγάλουμε και κάποιο αποτέλεσμα από τη χθεσινή και τη σημερινή συσκέψη θα ήταν πάρα πολύ θετικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστούμε κύριε Ευαγγελία Καρακώστα. Ε, και άλλη μια ερώτηση. Τελευταία ερώτηση από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, η κυρία Καταροβίτς. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη. Ε, ε, συγγνώμη. Λυπάμαι πάρα πολύ που η κυρία Βεζιά έχει φύγει από την ε, συνάντηση. Ήθελα να τη συγχαρώ. Διότι μας ε, έδειξε ότι έχουμε κοινέ αξίες όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ότι στο επίκεντρο της προσοχής μας βρίσκεται ο άνθρωπος κάθε άνθρωπος ε, και κυρίως οι χιλιάδες ε, αθώες γυναίκες και τα αθώα παιδιά που παίρνουν τη Μεσόγειο και χάνουν τις ζωές τους εκεί. Αυτή τη στιγμή είναι απίστευτο πως ορισμένες χώρες είναι έτοιμες να κλείσουν τα σύνορά τους και να απαγορεύσουν την είσοδο σε αυτούς τους ε, πρόσφυγες διότι κάθε ανθρωπινό έχει τα δικαιώματα του που ε, θεσπίζονται στην παγκοσμία διακήρυξη και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ε, πολύ καλή εντύπωση όταν ακούω τους συναδέλφους από χώρες που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ όπως η Ελλάδα, η Τουρκία, η Σερβία έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και για μένα είναι απίστευτο ότι ορισμένες χώρες βγαίνουν και λένε ότι δεν θα δεχθούν πρόσφυγες λόγω της θρησκείας τους. Με τρομάζει, διότι εγώ προερχόμαι από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, μια χώρα όπου ο πόλεμος σταμάτησε μεν πριν από 20 χρόνια, αλλά δεν έχουμε ξεχάσει τι συνέβη με τους πρόσφυγες και πόσο υποφέραμε πριν από 25 χρόνια. Αυτό που με ενισχύει ιδιαίτερα είναι ότι η εμπορία ανθρώπων αποτελεί μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι παλαιότερα. Όσον αφορά τις προσπάθειες τη Frontex, θα ήθελα να σας συγχαρώ ως ε, ε, διευθυντή μιας τέτοιας ε, οργάνωσης ε, για την εξαιρετική πρόοδο που έχει σημειωθεί και με τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ειδικότερα στις χώρες της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων. Και εγώ ως μέλος της Βοσνιακής Αντιπροσωπείας θα ήθελα να σας παροτρύνω να συνεχίσετε με το ίδιο εξαιρετικό τρόπο να κάνετε τη δουλειά σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη δήλωση αυτή. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας προχωρήσουμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι της συνεδρίασης το θέμα της ε, βελτιωμένης κοινοβουλευτικής ε, επίβλαψης ε, και την βελτίωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Να καλέσω τον κύριο Κεφαλογιάννη, Έλληνα μέλος του Κοινοβουλίου και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων είναι επίσης πρόεδρος ε, της ε, Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Κύριε Κεφαλογιάννη. Πρώτα απ' όλα θέλω να καλωσορίσω και εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλους τους συμμετέχοντες στην διακοινοβουλευτική διάσκεψη για το προσφυγικό και ακούγοντα πολλέ και εξαιρετικέ συγγύσει που έγιναν, θέλω να ξεκινήσω θετικά, γιατί συζητούμε ένα θέμα πολύ δύσκολο και για του ανθρώπου, αλλά για τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, Είναι ένα οργανισμό που μα εξασφάλισε 70 χρόνια ειρήνη και 70 χρόνια δημοκρατία για εμά τι χώρε του Ευρωπαϊκού Νότου, 40 χρόνια καλή δημοκρατία και όλες οι χώρες των Βαλκανίων αλλά και όλες όσες ζητούν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές τις δυο, αυτά τα δύο μεγάλα αγαθά θέλουν να εξασφαλίσουν. Και αυτή είναι και η μεγάλη πρόκληση που έχουμε για το μέλλον. Η Ευρώπη έκανε πάντα δύο βήματα μπρο και ένα πίσω, αν δει κανείς την ιστορία τη όλα αυτά τα χρόνια. Πάντα όμω έμεινε ένα βήμα να κάνει μπροστά. Δυστυχώ, στη σημερινή εποχή κάνουμε άλματα προ τα πίσω. Και αυτό το διαπιστώνουμε τώρα έχοντας δυο συν μία μεγάλες κρίσεις. Την οικονομική κρίση που βίωσε η Ευρώπη γιατί έχει κάνει βήματα πίσω, δεν προχώρησε στους θεσμούς της ολοκλήρωσής της και στον οικονομικό και στον πολιτικό τομέα και στο προσφυγικό που είναι το θέμα μας. Και έχουμε και μπροστά μας, θα το δούμε την Κυριακή, μια άλλη κρίση, ελπίζω πως όχι, με το ξύλωμα ενδεχομένω εισαγωγικά μια χώρα που είναι με το ένα πόδι μέσα και με το άλλο πόδι έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα τι διαπιστώνουμε. Διαπιστώνουμε ότι 70 χρόνια κάναμε αρκετά και σημαντικά βήματα στην οικονομία με την κοινή αγροτική πολιτική το 50 με το κοινό νόμισμα που προσπαθήσαμε να κάνουμε το 70 και δεν πετύχαμε με την κοινή αγορά που κάναμε το 90 με το ευρώ για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση αλλά δυστυχώ δεν κάναμε οικονομική νομισματική ένωση, δεν κάναμε ο ναι, κάναμε μόνο ναι, δηλαδή βάναμε μόνο την νομισματική ένωση και βρεθήκαμε σε ένα σημείο να μην έχουμε τα εργαλεία να αντιμετωπίσουμε τι κρίσει. Πολύ σύντομα θέλω να σα πω ότι η Ευρώπη βίωσε δραματικά την κρίση την οικονομική και κυρίω στι χώρε του Ευρωπαϊκού Νότου διότι δεν είχε τα εργαλεία που είχε η οικονομία των ΗΠΑ από την οποία ξεκίνησε και η κρίση έχει 6% του ακαθάριστου της εθνικού προϊόντος σε ομοσπονδιακό προϋπολογισμό και και την κρίση την οποία εξήγαγε στην Ευρώπη. Εμείς έχουμε το ένα. Δεν είχαμε τα εργαλεία τα πολιτικά. Ξεκινήσαμε εμείς μετά από τους παγκόσμιους πολέμους να κάνουμε πολιτική ολοκλήρωση. Θέλαμε τότε να κάνουμε την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση, European Defense Community. Και για δύο ψήφους στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση αυτή η πολιτική ολοκλήρωση δεν προχώρησε. Κάναμε την Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση που σήμερα τη χρειαζόμαστε, ένα θνησιγενή οργανισμό ο οποίο πέθανε στα μέσα τη δεκαετία του 90. Και σήμερα τι έχουμε, έχουμε ένα προπολογισμό όπω άκουσα των 100 εκατομμυρίων για τη φρόντε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι είναι 100 εκατομμύρια ευρώ, δύο ημερών τόκι του ελληνικού χρέου, το οποίο είναι 300 δισεκατομμύρια. Σε μια Ευρώπη που έχει χρέο 23 εκατομμύρια. Σημαίνει δηλαδή ότι δεν έχουμε τα εργαλεία να κάνουμε τη δουλειά μας. Έχουμε κι άλλο ένα εχθρό στην Ευρώπη. Είναι ότι συζητούμε πολύ και κάνουμε λίγο. Για κοιτάξτε τι κάναμε στο προσφυγικό. Η Ευρώπη δεν στάθηκε ικανή να διαχειριστεί ένα εκατομμύριο πρόσφυγες. Όταν χώρες όπως ο Λίβανος διαχειρίστηκαν ακόμα και σήμερα έχουν 1,2 εκατομμύρια πρόσφυγες στο έδαφος του, 25% του πληθυσμού τους. Και αντί η Ευρώπη να σκέφτεται με όρους μέλλοντος πώς θα σταθεροποιήσει μια δύσκολη πολιτική κατάσταση στο Λίβανο, φαντάζεστε να καταρρεύσει ο Λίβανος ως κυβέρνηση. Και αυτό το 1,5 εκατομμύριο του κόσμου να ψάχνει να βρει, το να ψάχνει να βρει διέξοδο στην Ευρώπη. Έχουμε την Ιορδανία, η οποία διαχειρίζεται 1,8 εκατομμύρια πρόσφυγες. Η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ιορδανίας είναι προσφυγούπολης. Με 80 εκατομμύρια πρόσφυγες. Έχουμε την Τουρκία, η οποία διαχειρίζεται 3 εκατομμύρια πρόσφυγες. Και δεν ξέρω και πόσοι άλλοι είναι μέσα στις διάφορες πόλεις μη καταγεγραμμένοι. Και η Ευρώπη δεν μπόρεσε να διαχειριστεί η Ευρώπη των αξιών, των αρχών, του πλούτου, μια από τις πιο προοδευμένες περιοχές του κόσμου ένα εκατομμύριο πρόσφυγες. Άρα έχουμε αποτύχει. Και πρέπει αυτό να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Γι' αυτό πέρα από το να συζητούμε και να κάνουμε διαπιστώσεις, στην Ευρώπη χρειαζόμαστε ηγεσία. Και δεν έχουμε ηγεσία. Πρέπει να κάνουμε να πάμε προς τα πίσω και να δούμε αυτοί οι οποίοι οραματίστηκαν την Ευρώπη μετά από εκατόμβες νεκρών, τι είδαν μπροστά και να πείσουμε και τον κόσμο. Διότι στην Ευρώπη σήμερα έχουμε φυγόκεντε δυνάμεις λαϊκισμού. Ο μεγάλος εχθρό του να λύσουμε αυτά τα προβλήματα είναι ο λαϊκισμός. Και λαϊκισμό έχουμε και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Δεν έχει χρώματα ούτε κόμματα ο λαϊκισμός. Στην Ευρώπη έχουμε το λαϊκισμό της Λεπέν στη Γαλλία, έχουμε το λαϊκισμό του Φάρετ στην Αγγλία, έχουμε το λαϊκισμό του Γκρίλο στην Ιταλία, έχουμε το λαϊκισμό, ελπίζω τώρα με τι νέε εκλογέ και τα νέα άρθρα που γράφει ο κύριος τον Ποδέμος να φύγει από αυτή την κατηγορία στην Ισπανία και είχαμε, έτσι ελπίζω, και το λαϊκισμό του Τσίπρα στην Ελλάδα το 2015, ελπίζω όχι τώρα. Και αν δεν κερδίσουμε τους λαϊκιστές, η Ευρώπη θα έχει φυγόκεντρε δυνάμεις. Και θα φτάσουμε πίσω, εκεί που θα χαθούμε κι εμείς οι ίδιοι. Άρα είναι κάτι που πρέπει να το δούμε προχωρώντας με γρήγορα βήματα μπροστά. Και εκεί αυτή τη μάχη πρέπει να την κερδίσουμε και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, έχουμε κάνει κάποιες συμφωνίες. Οι συμφωνίες αυτές πρέπει να πάρουν σάρκα και οστά. Δεν μπορεί, επειδή καταστρέψαμε τα ευρωπαϊκά σύνορα δηλαδή μεταφέραμε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν και τα σύνορα της Ελλάδας στην Ιδωμένη που είναι μια ύβρις για τις ευρωπαϊκές αξίες. Ύβρις. Δεν καταφέραμε εμείς οι Ευρωπαίοι παρά να κάνουμε αυτή την παρα... πα... παραγκούπολη η οποία ευτυχώ έκλεισε τώρα και μεταφέραμε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Σκόπια που τα Σκόπια ακριβώς γιατί ήθελαν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραβιάζοντας πολλές φορές και τις συνθήκες της Γενέβης έκλεισαν τον ευρωπαϊκό δρόμο και τώρα ναι, δεν έχουμε ροές στην Ελλάδα. Αλλά όλοι αυτοί οι απεγνωσμένοι άνθρωποι δεν θα ψάξουν να βρουν τους δρόμου τους μέσα από τη Μάλτα, από την Ιταλία ή από άλλους δρόμου. Όλοι αυτοί οι απελπισμένοι άνθρωποι της Ποσαχάριας Αφρικής που είναι εκατομμύρια εκατομμυρίων. Δεν θα ψάξουν να βρουν διέξοδο οι άλλοι απελπισμένοι από τρεις χώρες διαλυμένες, όπω είναι η Συρία, όπω είναι το Ιράκ, όπω είναι η Λιβύη, δεν θα ψάξουν να βρουν δρόμου. Άρα εμεί χρειαζόμαστε μια πολιτική συνεχτική, με αποφάσεις όχι γραφειοκρατικές και με προϋπολογισμό που μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ για την πρώτη συνάντηση που έγινε στη Μάλτα. Διότι το πρόβλημα δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε στα σύνορά μας. Το πρόβλημα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε κάνοντας ομόκεντρους κύκλους ανάπτυξης στις χώρες που έχουν τα προβλήματα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλούσια εμπειρία. Οι συμφωνίες ΛΟΜΕ, παραδείγματο χάρη, που είναι τον πρώην ε, οικονομικά ανθυρών κρατών με τις πρώην απικίες τους ήταν το 1964. Άρα έχουμε τα εργαλεία. Η κοινή αγροτική πολιτική ήταν μια, μια πολιτική επιδότησης της ευρωπαϊκής παραγωγής για να μην περάσουμε πείνα όπως περάσαμε στους παγκόσμιους πόλεμους. Άρα όλα αυτά πρέπει να τα δούμε με ανοιχτό μυαλό και με όρους μέλλοντος. Και όχι και εμείς οι πολιτικοί λαϊκίζοντας να περάσουμε τα επόμενα δύο χρόνια και τις επόμενες εκλογές. Υπάρχει ο χρόνος της πολιτικής, αλλά υπάρχει ο χρόνος της ιστορίας. Και εκεί που θα κρυθούμε είναι στην ιστορία. Το τι θα αφήσουμε πίσω μας, διότι όλοι θα κρυθούμε πολύ αυστηρά για αυτό που συμβαίνει. Ε, και σε ευρωπαϊκό και σε πολιτικό επίπεδο πρέπει να πάμε κόντρα στο ρεύμα. Διότι και σε εθνικό επίπεδο λαϊκίζομαι. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτά που συμβαίνουν για χώρες αλληπορημένες όπως είναι οι χώρες του Βίζεγκρατ. Που έζησαν και βίωσαν τον ολοκληρωτισμό. Και σήμερα φερόμενοι με ακραίες δράσεις ως θύτες οι ίδιοι. Μέσα από τα εθνικά κοινοβούλια υψώνουν τύχη. Εγώ πιστεύω ότι η Αυστρία έχει δώσει το μερτικό της συνεισφορά τη παίρνοντα 100.000 ή 80.000 πρόσφυγες όπως και η Σουηδία. Αλλά πρέπει αυτά να τα δούμε σε μια ευρωπαϊκή πολιτική η οποία θα μα δεσμεύει όλους. Ευρώπη αλλά καρτ δεν υπάρχει. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εμείς στο Κοινοβούλιο πρέπει να δώσουμε τη μάχη έβλεπα μια στατιστική πρόσφατη η οποία δείχνει απαντά στο ερώτημα αν συμφωνείτε με τον τρόπο αντιμετώπιση Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το προσφυγικό ζήτημα. Ξέρετε ποια είναι τα αποτελέσματα. Στην Ελλάδα είναι 94% ερευνητικέ απόψεις ενός λαού που είχε 80% υπέρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση διάθεση. Γιατί μιλήσαμε ζήσαμε δικτατορία όπω η Ισπανία και στην Πορτογαλία. 5% υπέρ. Στη Σουηδία την πιο ανοιχτή κοινωνία συμφωνεί με την πολιτική της Ευρωπαϊκής το 10% και διαφωνεί το 88%. Στην Ιταλία συμφωνεί το 17%, διαφωνεί το 77% και στην Ολλανδία ή στη Γερμανία το 26% και έχει αρνητική γνώμη το 67% και στην Ολλανδία που είναι μια άλλη φιλελεύθερη κοινωνία έχει αρνητική άποψη το 63% και συμφωνεί το 31%. Και όλες οι άλλες χώρες ανάμεσα σε αυτές. Χρειάζεται λοιπόν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια να δώσουμε αυτή τη μάχη. Αλλιώς μέσα στην παγκοσμιοποίηση η Ευρώπη κινδυνεύει να πάθει αυτό που έπαθε ο δεινόσαυρος. Επειδή δεν εξυγχρονίστηκε, εξαφανίστηκε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Μανώλης. Ευχαριστώ πολύ για τα πολύ ενδιαφέροντα σχόλιά σου. Ελπίζω ότι θα δρομολογηθεί μια σύντομη συζήτηση. Υπάρχουν ερωτήσεις ε, ή παρατηρήσεις από το κοινό. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Είμαι ε, Τούρκο Κοσοβάρα, βουλευτής. Νωρίτερα έγινε λόγος για, το, για τα κινήματα μεταναστών σε σχέση με το κοσμοπέδιο και την κατάσταση εκεί. Θα ήθελα εγώ προσωπικώς να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για την διοργάνωση της σημερινής συνεδρίασης η οποία, και χθεσινής η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη και σε ευχαριστώ πολύ. Χθες ήταν 20 Ιουνίου η Παγκόσμια ημέρα για τους πρόσφυγες. Βλέπουμε ότι πόσο μεγάλα είναι τα προβλήματα και τα νούμερα των προσφύγων και μεταναστών. Ε, ε, είναι ανεπαρκής, όμως οι λύσεις που προσφέρονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι μεγαλύτερη κοινότητα αξιών θα, περιοριστεί, θα περιοριστεί μόνο στα λόγια, δεν θα μπορέσει να δώσει απτές προτάσεις και λύσεις. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την επιβίωση μιας ολόκληρης γενεάς. Μέσα σε μια γενεά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συλλέξει εμπειρία που εάν δεν αξιοποιηθεί για να λύσει το μεταναστευτικό και προσφυγικό πρόβλημα, Νομίζω ότι, το ε, θα αποδειχθεί πως δεν έλειπαν τα χρήματα, αλλά η πολιτική βούληση. Υπάρχουν όλο και νέοι νόμοι για να μην μπορεί κανείς να μπει ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην μπορεί να ενταχθεί ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες βεβαίως δυσκολεύονται όλο και περισσότερο στην ε, διαδικασία ένταξης και οι πολίτες τους προσπαθούν ε, με άλλους τρόπους να μπουν στις χώρες Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν μπορούμε να μιλήσουμε διαρωτώμε για αποτυχία της μεταναστευτικής πολιτικής ή ιδιαιτέρως εάν κοιτάξουμε και την τελευταία φάση της συμφωνίας επανεισδοχής με την Τουρκία, εάν ε, εδώ έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν από τις χώρες τους για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για να τους αποτρέψουμε εμείς υψώνουμε φράκτες και σειρματοπλέγματα ή μήπω πρέπει και να ανοίξουμε πυρ τελικά γιατί ε, η τουρκική δημοκρατία θα πρέπει ε, να ε, μην εγκαταλειφθεί μόνη της μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Επανεισδοχής ε, στη διαχείριση του προβλήματος. Θα πρέπει νομίζω να σκεφτούν όλες οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρόβλημα αυτό σε όλους τους διαστάσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο αυτό. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο. Αν όχι, λέω να κάνουμε ένα διάλειμμα για καφέ. Θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για άτυπες συζητήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.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

Okay. Uh, Κυρίες και κύριοι, μετά από αυτό το σύντομο διάλειμμα, παρακαλώ, λίγη ησυχία. Ο κύριος Τζαμπάσκι θα μας κάνει μια παρουσίαση τώρα, που είναι μέλος ε, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ο οποίος είναι επίσης αντιπρόεδρος ε, της Αντιπροσωπείας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, την Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή και συμμετέχει σε πολλά ε, φόρα ε, που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών. Είναι ο κύριος ε, Τζαμπάσκι, ένας από τους πιο δραστήριους ευρωβουλευτές και πολλές φορές έχει τοποθετηθεί ως προς το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί εκπρόσωποι των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων. Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Αγαπητοί φίλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Εθνικών Κοινοβουλίων, των Κοινοβουλίων των Βαλκανικών κρατών, θέλω να αναφερθώ στην προηγούμενη τοποθέτηση του κυρίου Κεφαλογιάννη που αναφέρθηκε στο κοινοβουλευτικό έλεγχο και ιδιαίτερα την ε, υποχρέωση για διαφάνεια και λογοδοσία σε ένα δημοκρατικό σύστημα. Καθήκον των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι αυτή η επιτήρηση της λειτουργίας της εκτελεστικής εξουσίας, ο έλεγχος, η απόδοση λογαριασμών. Καλούν λοιπόν τα κοινοβούλια σε λογοδοσία της κυβερνήσεις. Και εξετάζουν και αν οι κυβερνήσεις έχουν δράση με βάση τις προσδοκίες και απαιτήσει της κοινωνίας. Είναι δηλαδή μια γέφυρα μεταξύ της κοινωνίας και των πολιτών τα κοινοβούλια και συμβάλλουν στον ε, κοινωνικό διάλογο σε διάφορα θέματα. Λυπούμε ιδιαιτέρως για το γεγονός ότι διαπιστώνω με λύπη μου όλο και περισσότερο πως τα κοινοβούλια δεν επιτελούν αυτό το έργο ή το επιτελούν όλο και λιγότερο και ε, εκπροσωπούν όλο και περισσότερο τις κυβερνήσεις του δρούν ω φερέφανο των κυβερνήσεων. Όλο και περισσότερο λοιπόν τα πολιτικά κόμματα επιδιώκουν την πλήρη επικράτηση με τις πλειοψηφίες στα κοινοβούλια έτσι ώστε οι ε, να έχουν απόλυτη εξουσία μέσα στις βουλές, αλλά ταυτόχρονα και μέσα από την κομματική πειθαρχία προσπαθούν να ελέγξουν τη συμπεριφορά των ε, κοινοβουλίων. Εγώ θα ήθελα να δώσω δύο σχετικά παραδείγματα. Καταρχάς από την ε, Βουλγαρία, το πολιτικό μου κόμμα είναι στον κυβερνητικό συνασπισμό της χώρας μου, αλλά και υποστηρίζουμε απλώς την κυβερνητική πλειοψηφία, χωρίς να έχουμε αναλάβει υπουργικού θόκους και έτσι υποστηρίζουμε την ε, κυβερνόσα πλειοψηφία εκφράζοντας τα συμφέροντα των ψηφοφόρων μας. Πολύ συχνά όμως διαπιστώνουμε ότι δεν λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των πολιτών από την κυβερνόσα πλειοψηφία. Αντίστοιχα το βλέπουμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό να λαμβάνονται υπόψη προς τώρα τα συμφέροντα των κρατών μελών και όχι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυπικά θεωρείται να είναι η κυβέρνηση της Ένωσης. Ασχολείται με την νομοθεσία, καταθέτει προτάσεις οι οποίες εγκρίνονται όχι γιατί είναι καλές τόσο, όσο γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χέρι της υποστήριξης της πλειονοψηφίας των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έτσι μπορεί να εξασφαλίσει τις ε, πλειοψηφίες που χρειάζεται για να εγκριθεί η πρότασή της. Αυτό το είδαμε πολύ πρόσφατα και σε μια συγκεκριμένη περίπτωση με μια πρόταση για τη Συμφωνία Άκτα η οποία είχε κινητοποιήσει ε, τους πολίτες. Οι πολίτες είχαν αντιδράσει πολύ έντονα στις προτάσεις Άκτα και ανάγκασαν έτσι τους βουλευτές να απορρίψουν τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο Κοινοβούλιο υπάρχουν πολλά κόμματα, εθνο, εθνικότητες, εκφράζονται διαφορετικές ομάδες πολιτών και συμφερόντων και έχουμε τη δυνατότητα έτσι να προβαίνουμε σε μια πολύ εντατική ανταλλαγή απόψεων και θέσεων. Πιστεύω ότι μπορούμε κατά αυτή την έννοια να αποτελέσουμε ε, υπόδειγμα για τα εθνικά κοινοβούλια. Πολλά είναι τα ζητήματα τα οποία ε, ανήκουν στο χώρο της επικουρικότητας, δηλαδή πρέπει να γίνεται η αντιμετώπιση του σε εθνικό επίπεδο, αλλά με συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων. Εγώ ως εισηγητής, ισκιώδης εισηγητής αντίστοιχα, συχνά έχω, συχνά έχω να κάνω με ερωτήσεις από διάφορες οργανώσεις πολιτών που μου ζητούν να υπερασπιστώ το δικαίωμά τους, τα δικαιώματά τους. Εμείς ως βουλευτές οφείλουμε να αφουγκραστούμε αυτές τις διαφορετικές ε, προτάσεις και θέσεις των πολιτών, ώστε να κάνουμε όσο καλύτερα τη δουλειά μας εκπροσωπώντας τους. Αυτό είναι το καθήκον μας. Να είμαστε ο διαμεσολαβητής μεταξύ του πολίτη και της εκτελεστικής εξουσίας με τις μεταναστευτικές ροές από την Ευρωπαϊκή Ένωση πέρσι είδαμε πόσο πιέστηκε το κάθε κράτος μέλος και πόσο σημαντικές ροές έφτασαν στα σύνορα των κρατών Αυτό ισχύει και για την Μακεδονία. Αυτός είναι ο ορισμός που εμείς επιλέγουμε. Πρόκειται για ένα μικρό κράτος με τεράστιες δυσκολίες λόγω αυτής της μεταναστευτικής πίεσης και της μεταναστευτικής κρίσης. Δυστυχώς όμως δεν γίνεται παρκός λόγος για τα αίτια των μεταναστευτικών ροών. Όπως επίσης δεν γίνεται παρκός λόγος για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες αυτών των αιτίων που είναι οι μακροχρόνιες συγκρούσεις και σειράξεις που προξενούν πάρα πολλά ανθρώπινα θύματα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξουν προτάσεις για την ε, ανακατανομή όπως λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας λέει ότι θα πρέπει να γίνει ανακατανομή των ε, προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα και την Ιταλία. Εδώ οι συμφωνίε έχουν υπογραφεί στη δεκαετία του 90 με τελείω διαφορετικέ συνθήκε μετανάστευση και προσφυγικού, αλλά και τελείω διαφορετική πολιτική κατάσταση. Πολιτικού πρόσφυγε βλέπαμε εκείνη την εποχή από το πρώην Ανατολικό μπλοκ. Έτσι λοιπόν η συμφωνία, η συμφωνία του Δουβλίνου δεν έχει σχεδιαστεί ώστε να αντιμετωπίσει τι τεράστιε πιέσει μεταναστευτικέ στα σύνορα τη Ελλάδα, τη Μακεδονία, τη Βουλγαρία. Μετά τη συμφωνία του Δουβλίνου, με βάση τη συμφωνία του Δουβλίνου, δεν μπορούν να καταγραφούν ε, ε, ε, εάν δεν κάνουν αίτηση για άσυλο, δεν μπορούν να παραμείνουν στην επικράτεια ενός κράτους οι πρόσφυγες. Τα εθνικά κοινοβούλια λοιπόν θα πρέπει να συνεργαστούν περισσότερο στη διαδικασία για την αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας το Εθνικό Κοινοβούλιο στην Ελλάδα Φερρυπίν ξέρει πολύ καλύτερα από τον καθένα ποια είναι η κατάσταση και ξέρει και καλύτερα από τον καθένα τι γνώμη έχει ο ελληνικός λαός για το πώς θέλει να αντιμετωπιστεί η κρίση. Κατά τη λήψη των αποφάσεων, λοιπόν, κατά, την, ε, κατά τον προσδιορισμό των πολιτικών επιλογών στο τομέα αυτών, δεν λαμβάνονται παρκώ υπόψη τα συμφέροντα των πολιτών. Και ιδιαίτερα θέλουμε να τονίσουμε πως η μεταναστευτική πολιτική ε, έχει μετατραπεί τελικά σε μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ των χαρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και των χαρών της δυτικής Ευρώπης, εκείνων που θεωρούνται ίσως εξωτερικά σύνορα και εκείνων ε, που ε, πλήττονται από τα ρεύματα μετανάστευσης. Οι προτάσεις Επιτροπής έχουν παραμείνει επί χάρτου μόνο, δεν έχουν προχωρήσει και είναι όλο και περισσότερο, όλο και μεγαλύτερο το πρόβλημα και ιδιαίτερα για τις χώρες οι οποίες είναι υποψήφιες για ένταξη. Υποστηρίζω τις προσπάθειες για την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων και των ελέγχων και επίσης υποστηρίζω τις προτάσεις για βελτίωση της ποιότητας ζωής και, την, και για την κατάργηση, απάλληψη των λόγων που οδηγούν στην παράτυπη μετανάστευση. Πρέπει λοιπόν να απαλληφθούν οι λόγοι που οθούν του ανθρώπου στη μετανάστευση και αυτό είναι το βασικό που έχω να πω. Όλα τα, όλα υπόλοιπα είναι μόνο παρηγορητικά μέσα και δεν δίνουν απάντηση στο πρόβλημα. Δεν μπορούμε φυσικά να, πάρουμε, να υποδεχθούμε όλους τους πρόσφυγες από τη Μέση Ανατολή, το Αφγανιστάν, το Ιράν και ε, όλες τις άλλες χώρες που έχουν προβλήματα. Οι χώρες των Βαλκανίων βρέθηκαν ε, στην πρώτη γραμμή υποδοχής των μεταναστευτικών ρευμάτων, κυρίε και κύριοι. και πλήγησαν και από ε, δηλώσεις που έγιναν ε, ελαφρά την καρδία και χωρίς ε, περαιτέρω περίσκεψη από ηγετικές μορφές των κρατών της Δυτικής Ευρώπης όπως ε, της ε, καγκελαρίου Μέρκελ ή του Προέδρου Ολόντ. Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσφέρει για να υποστηρίξει τα κράτη αυτά και οικονομική βοήθεια αλλά πάνω απ' όλα μακροπρόθεσμες λύσεις και πιστεύω ότι οι συνομιλίες μέσα στα κοινοβούλια είναι ένα μέσον καλό, όπως είπα και νωρίτερα και η πολιτική μου ομάδα ECR, συντηρητικοί μεταρρυθμιστές της Ευρώπης και εγώ προσωπικώς υποστηρίζουμε μια διαφορετική πολιτική μετανάστευσης και ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εν μέρει υποστηρίζει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι πρέπει να ε, εργαστούμε έτσι ώστε να μειωθούν οι μεταναστευτικές ροές, να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση των πολιτών και αυτό σημαίνει πως πρέπει να ενισχύσουμε τους ελέγχους στα σύνορα και να συνάψουμε περισσότερες συμφωνίες επανεισδοχής, αλλά και να τις εφαρμόσουμε και να μην αρκούμεθα μόνο στο να προσφέρουμε οικονομική ενίσχυση για τους πρόσφυγες. Βλέπω όμως ότι δεν συμβαίνει αυτό στην πράξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ε, προβαίνει σε μεμονωμένες δράσεις και μέτρα και αντί να φροντίσει να εξασφαλίσει ηρεμία και ασφάλεια με τις ε, απερίσκεπτες κινήσεις της, με τις απρογραμμάτιστες, ασχεδίαστες κινήσεις της η Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγεί σε όλο και περισσότερα προβλήματα. Για το συνάλφο γιατί στην Σίνικ από το κοσφοπέδιο του Κοσφοπεδίου που μίλησε για την Τουρκία και την πολιτική της, θα ήθελα να απαντήσω τα εξή. Έχουμε πολλά εκκρεμή ζητήματα σε σχέση με την Τουρκία και την πολιτική της. Έχουμε μια μη λογική δραστηριότητα και πράξη του Τούρκου Προέδρου σε σχέση με την ασταυτική πολιτική γιατί την αξιοποίησε για να εκβιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συμφωνίες επανεισδοχής δεν υλοποιούνται και δεν βλέπουμε από πλευράς της Τουρκίας καμία βούληση για τήρηση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει. Εγώ προσωπικώς Είμαι πολύ επιφυλακτικός σε σχέση με την ε, υλοποίηση της συμφωνίας αυτής με την Τουρκία. Νομίζω ότι προσπαθεί μόνο να κερδίσει χρόνο και χρησιμοποιεί τους μετανάστες και τις ροές μεταναστευτικές μόνο για να ασκήσει πολιτική ε, πίεση και να κερδίσει σε πολιτικό επίπεδο στο ιστορικό της χώρας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Τζαμπάσκι για την παρουσία σας εδώ σήμερα προκειμένου να συζητήσουμε αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πριν από δύο εβδομάδες παρεμπιπτόνως ε, η Μονάδα Δράσης η Προενταξιακή οργάνωσε μία διάσκεψη για την δράση των πολιτικών ομάδων και των κομμάτων ε, στην προενταξιακή διαδικασία και είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τους ομιλητέ να αναφέρονται σε διάφορες πτυχέ κοινοβουλευτικής δράσης, το ρόλο, τι ευθύνε τους, ε, προκειμένου να ε, συν να συντονίσουν τους διάφορες ε, εταίρους για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι η διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σήμερα μας μιλήσατε για το ποια θα πρέπει να είναι η απάντησή μας στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα σχόλιά σας. Θα ήθελα τώρα να κηρύξω ε, την έναρξη της συζήτησης ε, ο προσκεκλημένος μας από την Τουρκία. Παρακαλώ. Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συναδελφοί, ο κύριος Τζαμπάσκι από την ε, Βουλγαρία κατηγόρησε άδικα τον πρόεδρό μας και την πατρίδα μας και πρέπει να δώσω απάντηση. Ο κύριος πρόεδρος της Τουρκίας και η χώρα μας έχουν υποδεχθεί, όπως είπαμε και νωρίτερα, τρία εκατομμύρια πρόσφυγες και τους έχουν προσφέρει άσυλο. Με πάνω από 10 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια πρέπει να εννοεί ο μιλητής, ευρώ κόστος για την υποδοχή και την ε, στέγασή τους. Έτσι λοιπόν η Τουρκία με 80 εκατομμύρια ε, πληθυσμό και 10.000 κατακεφαλήν εισόδημα έχει υποδεχθεί 3 εκατομμύρια πρόσφυγες. Αυτή τη στιγμή στις ακτές του Αιγαίου έχουμε πάνω από 10.000 πρόσφυγες, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους ε, που πνίγηκαν προσπαθώντας να περάσουν στις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανείς δεν τα λέει αυτά. Το... Ο, ο δε κύριος πρόεδρος της Τουρκίας το μόνο που ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να επιτελέσει τις ανελημμένες υποχρεώσεις της. Ούτε εκβιασμός υπήρξε, ούτε είναι δυνατόν να δεχθούμε τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς. Ας δούμε λοιπόν το, η Βουλγαρία πόσους ε, πρόσφυγες έχει υποδεχθεί και πόσες ε, δαπάνες έχει επιβαρυνθεί για την υποδοχή τους. Ας το δούμε αυτό για να συζητήσουμε σε ε, ανοιχτούς όρους. Εμείς ε, σας καλούμε να έρθετε στους καταβλισμούς, να τους επισκεφθείτε, να δείτε τις συνθήκες που έχουμε εξασφαλίσει για την ε, διαμονή των προσφύγων. Είναι σαν να είναι δικοί μας η ποιότητα της ζωής που τους προσφέρουμε. Και ως εκ τούτου θέλω να πω ότι καταδικάζω και απορρίπτω τα λόγια που ακούστηκαν. Uh, uh, Θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε. Τώρα βλέπω ότι γίνεται έτσι μια θερμή συζήτηση. Κύριε Τζαμπάσκι, έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητές συνάδελφε. Ελπίζω να μην θεωρείτε ότι θίγεστε προσωπικά από αυτή την πολιτική μου αξιολόγηση. Λυπούμε ιδιαίτερως αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά θα σας καλέσω και εγώ να έρθετε στα τουρκοβουλγαρικά σύνορα και να δείτε πώς περνούν με λεωφορεία αλλά και με άλλα οχήματα μέσα από την πράσινη γραμμή οι μετανάστες χωρίς να τους ελέγξουν ή να τους περιορίσουν σύνοριοφύλακες από πλευράς τουρκικής. Υπάρχει συμφωνία επανεισδοχή, επαναπροώθησης μάλλον μεταξύ τουρκική και βουλγαρικής δημοκρατία, αλλά δεν τηρείται αυτή. γιατί δεν έχει του ίδιου όρου με αυτό είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη Συμφωνία ευρωπαικη Ευρωπαϊκή Ένωση-Τουρκία. Έχουμε λοιπόν πολλού οι οποίοι έχουν περάσει παράτυπα από τα σύνορα τη Τουρκία στο βουλγαρικό Έδαφο. Μα ανησυχεί ιδιαίτερα το πρόβλημα αυτό, είναι σοβαρό πρόβλημα. Γι' αυτό και σα καλώ να έρθετε στα δικά μα σύνορα για να δείτε την κατάσταση με τα μάτια σας. Ευχαριστούμε. Τώρα ο Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου της ε, πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, ο κύριος Ραφή Σαρίτη. Έχετε το λόγο. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μια ένωση αντιπροέδρων, ναι, παρεπιπτόντως per integrim në Republikën e Maqedonisë, që do të thotë nga komuniteti shqiptar. No translation, not yet. Ένα λεπτάκι μόνο γιατί κάποιο κουμπί δεν πατήθηκε σωστά, μα συγχωρείτε. Can you continue? Είχε περάσει από το λάθος κανάλι μας, ακούτε τώρα. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι βουλευτής της Δημοκρατικής Ένωσης ε, για την ε, ένταξη και ανήκω στην αλβανική κοινότητα. Ζω στην ε, πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και θα ήθελα να είμαι πολύ ειλικρινής, χωρίς δημαγωγία, γιατί ακόμη και χθες και σήμερα ακούσαμε πολλές συζητήσεις, πολλά καλά λόγια, Και σε αυτή την αίθουσα γίνεται πολιτική σε μεγάλο βαθμό. Το λέω αυτό διότι ελθεύει και τονίστηκε από τους προλαλήσαντες ότι τα κράτη, τα βαλκανικά κράτη αποτελούν ε, κομμάτι μιας οδού διέλευσης ε, για πρόσφυγες από την Αφρική και από κάποια μέρη της ε, Μέσης Ανατολής. Ο προκάτοχός μου, ο, ο, βούλγαρος συνάδελφος που μόλις μίλησε, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι υποστηρίζει τη διατήρηση των συνόρων ταυτόχρονα με την τήρηση των, του επίπεδου που απαιτείται για τους πρόσφυγες παρότι ήταν κάπως αντιφατική η δήλωσή του το λέω αυτό διότι ο καθένας μας θα πρέπει να θεωρεί τη χώρα του, την οικογένειά του, τον εαυτό του υπό το πρίσμα του τι έχει κάνει για τους πρόσφυγες. Θα πρέπει λοιπόν να το κάνει ο ίδιος αυτό πριν επικρίνει τους άλλους. Το λέω αυτό διότι εγώ ο ίδιος ε, έχω φιλοξενήσει στο σπίτι μου πρόσφυγες ε, από τη Βοσνία το 1994, από το Κωσυφοπαίδιο. Τους έχω φιλοξενήσει στο σπίτι μου, στο χωριό όπου ζω. Λέτε όμως ότι πρέπει να διατηρήσουμε τα σύνορα, να προφυλάξουμε τα σύνορα. Ναι, αλλά σε ποια έκταση ώστε να πάψουν να χάνουν τις ζωές τους ε, πρόσφυγες στα σύνορα. Να σας υπενθυμίσω τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εμείς ε, ως Βαλκανική χώρα στο πρόσωπο ενός πρόσφυγα είναι ζωγραφισμένα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αλλά όχι όλα. Δεν λέω λοιπόν ότι δεν πρέπει να γίνεται ο σωστός έλεγχος, αλλά πρέπει να ξέρουμε τι όθησε τον κάθε άνθρωπο να αποφασίσει να μεταναστεύσει. Άλλοι για οικονομικούς, άλλοι για άλλους λόγους. Αλλά θα ήθελα να επαναλάβω ότι Καλό θα ήταν να είχαμε εδώ και κάποιον εκπρόσωπο από μια χώρα που έχει φιλοξενήσει ε, πρόσφυγες όπως ε, τη Γερμανία, τη Σουηδία. Καλό είναι που έχουμε εκπροσώπους της Ελλάδας, διότι η Ελλάδα έχει συμβάλει σημαντικά στην προστασία των προσφύγων. Κατά την άποψή μου δεν μπορούμε να επικρίνουμε ούτε την Τουρκία, διότι η συμβολή της Τουρκίας αυτή τη στιγμή όπως και της Γερμανίας. Ελάχιστες χώρες ε, έχουν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο προστασίας όπως αυτή προσφέρει η Τουρκία και η Γερμανία. Ακόμη και αν διαφωνείτε μαζί μου, έχω την εντύπωση ότι μπορείτε να καταλάβετε τι εννοούμε και ε, το να λέτε ότι εμείς ε, οι χώρες της Βαλκανικής έχουμε ε, κάνει ακραίες πολιτικές όσον αφορά τους πρόσφυγες και προσπαθούμε να φτιάξουμε δικές μας πολιτικές ε, που αντιβαίνουν των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να απαντήσω ότι ο καθένας μας θα πρέπει να δει τι κάνει ο ίδιος για τους πρόσφυγες, τι κάνει η Φιρόμ, τι κάνει η Βουλγαρία, τι κάνει το Μαυροβούνιο, τι κάνει η Αλβανία, όλες οι χώρες πόσο καλά είμαστε εξοπλισμένοι για να υποδεχθούμε τέτοιους ε, πρόσφυγες. Η απάντηση είναι ότι δεν έχουμε κάνει όσο θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει. Και κλείνω την ομιλία μου λέγοντας ότι δεν είναι εύκολο να υποδεχθεί κανείς πρόσφυγες ε, και στη δική μας χώρα. Διότι πρέπει να τους παρέχουμε υπηρεσίες κάποιου επίπεδου αλλά ξέρετε τα πρότυπα που έχουμε για μας είναι τόσο χαμηλά που είναι δύσκολο να έχουμε αντίστοιχες υπηρεσίες στους πρόσφυγες. Οι χώρες μας, οι πολιτικές μας ε, αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο ανθρωπιστικές λοιπόν που το λέω διότι κάποιοι προσπαθούν να αποκομίσουν όφελος από τη δυστυχία των προσφύγων αντί να τους υποστηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν να βρουν καταφύγιο. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα έπρεπε να είμαστε ικανοποιημένοι που ε, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ειρήνη στις χώρες μας ενώ μένεται πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αυτέ είναι οι συνθήκε που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα. Και έχουμε διάφορε χώρε που άμεσα ή έμεσα έχουν ασχοληθούν με το ζήτημα των προσφύγων και πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο για περισσότερη δράση. Ε, τέλος, θα ήθελα να πω ότι η δήλωσή σα ήταν πολύ σωστή και συμφωνώ μαζί σα αν μη τι άλλο, για τους ε, Βαλκανικού λαούς όπου τα κοινοβούλια εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις κυβερνήσεις μας. Εμείς ε, τα κοινοβούλια των Βαλκανικών χωρών ε, υπηρετούμε τις κυβερνήσεις μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Ε, ενώ σύμφωνα με το Σύνταγμα οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να, να έχουν λογοδοσία ως προς το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ραφή Σαλική. Ο κύριος Αλιόσκαγια. Από το Τουρκικό Κοινοβούλιο. I'm sorry, I'm sorry. From Turkish Parliament, Uh, uh, uh, <laughs> Κύριε Mr. ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δύο μέρες τώρα συζητούμε διεξοδικά το θέμα αυτό και προσπαθούμε να διατυπώσουμε με την καλή πρόθεση πάντα, με την καλή διάθεση συγκεκριμένες προτάσεις μας ικανοποιεί ιδιαίτερα σε αυτή η κατάσταση. Θα ήθελα λοιπόν να σημειώσω ότι βεβαίως τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να συμβάλλουν με τις προτάσεις τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αναμφίβολα. Και να εκφράσουν βέβαια πολιτική βούληση, η οποία θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και σε επίπεδο κυβερνήσεων και να μεταφράζεται σε απτές πράξεις. Έτσι λοιπόν, μαζί με τους βουλευτές μπορούμε να έχουμε μία ε, διακυβέρνηση ε, από πλευράς της κυβέρνησης πολύ πιο συγκεκριμένη, πιο αποτελεσματική, με συγκεκριμένα λύσεις και αποτελέσματα. Σε αυτό νομίζω ότι συμφωνούμε. Είναι διαφορετικές οι και οι προσεγγίσεις βεβαίως εμείς βλέπουμε ότι στην Τουρκία το πρόβλημα έχει πάνω απ' όλα ανθρωπιστικές διαστάσεις και αυτή είναι η πολιτική βούλαση με την οποία το προσεγγίζουμε στην Τουρκία. Βεβαίως, πρέπει να υπάρξει μια ταχύτερη αντιμετώπιση και πιστεύουμε ότι σε αυτό πρέπει να εργαστούμε περισσότερο στην Τουρκία, μια ταχύτερη αντιμετώπιση, πιο αποφασιστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Τώρα, στα όσα είπε ο κύριος Τζαμπάτσκι για την Τουρκία και την ε, κυβέρνησή της, ε, το μόνο που μπορώ να απαντήσω ήταν πολύ ατυχής οι παρατηρήσει. Έχουμε συζητήσει εδώ και δύο μέρες, έχουμε ακούσει τους εκπροσώπους όλων των κρατών που μίλησαν με επενετικά λόγια για τις προσπάθειες της Τουρκίας, για, ε, για την υποδοχή, για την ποιότητα της υποδοχής. Αυτό έχει καταγραφεί από όλου. και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να περιγράψει την κατάσταση με τα χρώματα του κ. Τσαμπάτσκι. Επίσης ε, και οι υπεύθυνοι που μίλησαν νωρίτερα για τι ε, συμφωνίε επανεισδοχής εξήγησαν ποια είναι η κατάσταση, ποιες είναι οι συνθήκες της παράτυπης μετανάστευσης και κινήσεις των παράτυπων μεταναστών ε, στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιες είναι οι συμφωνίες και οι, ε, τα μέτρα που εφαρμόζει η Τουρκία. Τώρα τον ισχυρίζεται κανείς ότι είναι ζήτημα είτε εκβιασμού, είτε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο η Τουρκία ε, στη διαπραγμάτευση για άλλα ζητήματα μέσα από τη Συμφωνία Επανεισδοχής, μου φαίνεται απολύτως ατυχής και ασφαλμένη εκτίμηση. Η Τουρκία έχει έναντι ολόκληρη της ε, ανθρωπότητας, της εθνούς κοινότητας και των ε, κρατών του κόσμου με ειλικρίνεια θέσει το ζήτημα το προσφυγικό, το μεταναστευτικό. Βεβαίως έχει πολύ μεγάλη σημασία η εθνική ασφάλεια, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να δώσουμε φωνή και να ακούσουμε και να προστατέψουμε την ψυχή μας και τη συνείδησή μας. Εάν αυτό δεν κοιτάξουμε, εάν δεν κοιτάξουμε την ανθρωπιστική μας υποχρέωση δηλαδή, τα έχουμε χάσει όλα. Αυτή είναι η δική μας η προσπάθεια να επιτελέσουμε το ανθρωπιστικό μας έργο. Και πιστεύω ότι σε αυτό θα πρέπει η κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κοιταχτεί στον καθρέφτη και να δει εάν η συνείδησή της της λέει πως έχει κάνει αυτό που όφιλε να πράξει στο έπακρον, όπως εμείς. Εμείς δεν δεχόμαστε να αξιολογηθούν οι προσπάθειες μας και οι συνομιλίες μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εκβιασμός. Έχουμε σχέσεις στρατηγικού επίπεδου και στρατηγικής πνοής με την Ευρωπαϊκή Ένωση 50 χρόνια τώρα δεν έχουμε να κάνουμε με σχέσεις, δεν πρόκειται για σχέσεις ενός ε, ανώτερου ή κατώτερου γραφειοκράτη υπαλλήλου. Δεν μπορούμε να πούμε ότι περιοδος αυτό. Είναι υψη του επίπεδου και στρατηγικής αξίας αυτές οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν καλό θα είναι και αντί να κοιτάμε δηλώσεις, να κοιτάμε καλύτερα τις πράξεις και μετά αφού κοιτάξουμε τι έχει πραγματικά γίνει στην πράξη και μπορέσουμε να έρθουμε αντιμέτωποι με τη συνείδησή μας, τότε μόνο μπορούμε να κάνουμε αξιολογήσεις τέτοιου τύπου. Ευχαριστώ πολύ. Thank you much indeed. Uh... Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο? Uh, okay. Uh, no answer. Okay. More quiet. Okay. Thank you. Maybe a good solution. Αγαπητοί συνάδελφοι, πλησιάζουμε στο τέλος ε, της ε, διήμερης ε, συνεδρίασής μας. Θέλαμε επίσης ε, να συζητήσουμε το θέμα της περιφερειακής συνεργασίας, της στενότερης συνεργασίας ε, και είναι εδώ η κυρία Γκόμες για να ε, μας μιλήσει γι' αυτό, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, μια ε, που είναι εδώ από το 2004, έχει τεράστια εμπειρία και ελπίζω ότι ο καλός μου φίλος, ε, ο φίλος μου ε, κύριος Κούκαν ε, θα δεχθεί να προεδρεύσει αυτό το τμήμα της συνεδρίασης. Ελπίζω να είναι επικοδομητική η συζήτησή μας. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ να αναλάβετε την Προεδρία. Distinguished ladies and gentlemen, good afternoon. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι Μεγάλη τιμή και χαρά για μένα να βρίσκομαι εδώ στη θέση του κυρίου Τσανέσκη και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος ε, γιατί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση θα δώσω ε, στην αξιότιμη συνάδελφο την ε, κυρία Γκόμες το λόγο που θα μας κάνει μια παρουσίαση για την ενίσχυση της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας και της περιφερειακής συνεργασίας των αρμοδίων αρχών. Άννα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά για μένα να βρίσκομαι ε, εδώ με τους συναδέλφους από διάφορα εθνικά κοινοβούλια. Ε, θα ήθελα και εγώ να ήμουν περισσότερο παρούσα κατά τη διάρκεια της ε, συνεδρίασης αυτής. Ε, και ελπίζω, ήλπιζα και άλλοι συναδέλφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετείχαν, ε, γιατί αυτός είναι ο τρόπος να προχωρήσουμε, να βρούμε σημεία επί των οποίων διαφωνούμε, αλλά σημεία επί των οποίων συμφωνούμε για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Πραγματικά, τη γνώμη μου, ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι ε, κρίσιμος ε, όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις σαν αυτές που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ε, ενδεχομένως να σας συγκλονίσω σε κάποια πράγματα που θα σας πω. αλλά πριν γίνω ευρωβουλευτής ε, ήμουν ε, διπλωμάτης ε, και χρειάστηκε να κρατάω το στόμα μου κλείστο. τώρα όμως που είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορώ πια να μιλάω και να εκφράζω την άποψή μου ανοιχτά. Λοιπόν, έχουμε την, ευθύνη να μην καταπίνουμε αμάση το οτιδήποτε μας λένε άλλοι και να, είμαστε, να σεβόμαστε την ε, εντολή ε, που έχουμε λάβει που είναι να επιβλέπουμε, να παρακολουθούμε την ε, εκτελεστική εξουσία για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στις αξίες που αναφέρονται στο Σύνταγμα των χωρών μας όμως επίσης και στις συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλους όσους είναι ήδη μέλη της Ένωσης αλλά και για όσους είναι στην προενταξιακή διαδικασία. Πιστεύω λοιπόν ότι υπήρξε κάποιο είδου έλλειμμα και γι' αυτό εγώ επικροτώ την ανταλλαγή ε, απόψεων τη σημερινή και ελπίζω να υπάρξει να υπάρξει συνέχεια. Γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, ειδικότερα τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών ε, που είναι στην πρώτη γραμμή της υποδοχής των μεταναστών, ε, μπορούν να δουν καλύτερα κάποια πράγματα, τα οποία εμείς εδώ από τις Βρυξέλλες πιο δύσκολα τα βλέπουμε και νομίζω ότι εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε το τεράστιο πλεονέκτημα να μπορούμε να ταξιδεύουμε. Έχουμε πάει ε, στην Τουρκία, στην Ελλάδα, ε, ναι, έχω πάει στο Λίβανο, στην Ιορδανία, στη Συρία πριν από τον πόλεμο ε, και μετά από τον πόλεμο. Ε, πήγα στη Λιβύη και σε πολλές άλλες χώρες και όχι μόνο εγώ αλλά και άλλοι πολλοί συνάδελφοι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω λοιπόν και επειδή είμαι και μέλος της Υποεπιτροπής Ασφάλειας ε, και Άμυνας, κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής μου εργασίας έχω ε, προσπαθήσει να διασυνδέσω τα ανθρώπινα δικαιώματα με την ασφάλεια ε, και την άμυνα. Είμαι κάποιος λοιπόν, ε, που είμαι ένας άνθρωπος που είναι πραγματικά πολύ ευαίσθητο σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγοι, οι πρόσφυγες δεν είναι αυτοί που μας απειλούν σε επίπεδο ασφαλείας. Καθόλου όσον αφορά την τρομοκρατία πολλές φορές επικρίνουμε τι ίδιε μα τι κυβερνήσει που μιλούν για του ξένου ξένους μαχητές, αλλά αυτοί που μας επιτίθενται είναι δικοί μας πολίτες. Πολίτες της Ένωσης. Είναι λοιπόν γελίο να μιλάμε για ξένους μαχητές όταν οι ίδιοι υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Μα επιτίθενται και πολλέ από τις πολιτικές μας εξηγούν για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, κυρίω από πλευρά των νέων. Λοιπόν, εγώ δεν ε, δέχομαι αυτούς που στιγματίζουν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, που θεωρούν ότι αυτοί ε, είναι υπεύθυνοι, είναι ο κίνδυνος ε, και η απειλή στην ασφάλεια μας. Ε, όπως ε, έχω πει, ο ευκολότερος τρόπος ε, είναι μέσω αυτών που ήδη επιχειρούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατά τη γνώμη μου δεν είναι μόνο μια κρίση προσφυγική, είναι μια κρίση δική μας Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν έχουμε ε, σταθεί στο ύψος των αξιών μας και αν δεν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις βασικές αιτίες ε, αυτής της ε, μετακίνησης των ανθρώπων, αν έχει να κάνει με την παγκοσμιοποίηση. Ναι, έχει. Έχει πάρα πολλές θετικές πτυχές, αλλά και πολλές αρνητικές η παγκοσμιοποίηση. Χρειαζόμαστε την κινητικότητα του κόσμου και οι άνθρωποι θέλουν πράγματι ε, να βελτιωθούν ε, και να βελτιώσουν τη ζωή τους. Ή, αν λοιπόν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό ε, στη χώρα σου, θα πας σε μια άλλη χώρα. Αυτή είναι η ιστορία της Ευρώπης. Εγώ είμαι Πορτογαλίδα, είναι η ιστορία της δικής μου της χώρας που έχει εξαγάγει πολύ κόσμο σε ολόκληρο τον κόσμο, ειδικότερα κατά τα τελευταία χρόνια με τις πολιτικές ε, λιτότητας. Να μην σας πω ότι αυτή τη φορά η εξαγωγή ανθρώπων ε, είναι διαρροή εγκεφάλων. Πάρα πολύ ε, εκπαιδευμένους ανθρώπους εξάγουμε πλέον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το θύμα της ίδιας της επιτυχίας, για να το πω έτσι. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και σε άλλα μέρη του κόσμου. Ε, όταν είναι ένας χώρος βελτίωσης του βιωτικού επίπεδου. Για ποιο λόγο να μην έρθουν ε, στην ε, Ευρώπη. Δεν θέλω να πάνε σε Σαουδική Αραβία προφανώς. Θέλουν να πάνε σε ένα χώρο που τους δίνει τις συνθήκες να μπορέσουν να ευημερήσουν και σε προσωπικό και σε οικογενειακό επίπεδο. Παράλληλα, η Ευρώπη είναι πάρα πολύ μικρή έχουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τη μικρότερη Ευρώπης, τη λιγότερη Ευρώπης, γιατί δεν έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε τις βασικές αιτίε ε, για, τους, για τις οποίες μίλησε ο κύριος Τζαμπάσκι και πολλοί άλλοι. Όλοι μιλάνε για αυτές τις ε, αιτίε. Ε, η εξωτερική μας ε, ε, ε, πολιτική, για παράδειγμα. Δεν τη χρησιμοποιήσαμε σωστά για να αποφύγουμε την σύγκρουση στη Συρία. Δεν είμαστε μόνοι βέβαια. Θα ήθελα η Ευρώπη να ήταν πιο ενεργός στην προσπάθεια αντιμετώπισης της σύγκρουσης της Συρίας. Η Λιβύη είναι μία ακόμη τέτοιου είδους περίπτωση, γιατί κατά τη γνώμη μου, και εγώ ήμουν εισηγήτρια για τη Λιβύη, πήγα εν μέσω πολέμου πολλές φορές και ξέρω ότι το πρόβλημα δεν ήταν η παρέμβαση παρέμβαση, τι δεν συνέβη μετά ήταν το πρόβλημα. Έχει τεράστια ευθύνη, ευθύνη η Ευρώπη ως προς αυτό, ειδικότερα ως προς την ανάπτυξη υποδομών, την ασφάλεια, την άμυνα κλπ η Λιβύη δεν είναι, ένας δεν είναι μια, μια χώρα που εξάγει ανθρώπους, είναι ένα μέρος το οποίο ε, εισέρεαν άνθρωποι από διάφορα μέρη του κόσμου και δεν νομίζω ότι ο τρόπος να το λύσει το πρόβλημα η Ευρώπη είναι η εξωτερική ανάθεση είτε στην Τουρκία ε, ε, ε, οπουδήποτε αλλού. Ε, το γεγονός δηλαδή ότι επικαλούμαστε τώρα τις δηλώσεις, τη δήλωση, τη συμφωνία με την Τουρκία. Δεν μπορούμε λοιπόν να πετάμε το μπαλάκι σε άλλες χώρες. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούμε πρόσφυγες και μετανάστες. Σκεφτείτε για παράδειγμα την Ερυθρέα, την Αιθιοπία, παρά το γεγονός ότι όλος ο κόσμος θεωρεί ότι η Αιθιοπία οποία έχει ένα καλό καθεστώ Όχι, είναι ένα κατασταλτικό καθεστώς. Να μην μιλήσω για το Σουδάν και για άλλα μέρη του κόσμου που ο κόσμος φεύγει για να σωθεί. Όπως είναι η περίπτωση της Νιγηρίας, για παράδειγμα, με το πρόβλημα του Μπόκο Χαράμ. Οπότε εμείς ε, είμαστε πραγματικά ε, το θύμα της ίδιας μας της ε, ε, επιτυχίας και πολύ λίγα κάνουμε για να μπορέσουμε να λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα το αποτέλεσμα λοιπόν είναι μια διαδικασία που ε, είναι καταστροφική ε, και δεν λύνει το πρόβλημα. Πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ χωρών όπου υπάρχουν σοβαρές προσπάθειες αντιμετώπισης προβλημάτων και ε, καθεστώτων που δεν είναι ασφαλή. Και έχουμε και πάλι μια τεράστια ευθύνη από αυτού, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι κάποια από αυτά τα καθεστώτα, ε, τα οποία καταχρώνται τους πόρους ε, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη των λαών τους, ε, το ενισχύουν αυτό μέσω διαδικασιών που περνούν και μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε τεράστια ευθύνη μας και εν προκειμένου. Τώρα, το η αποδοχή ότι η Ευρώπη χρειάζεται μετανάστες και πρόσφυγες. Χρειάζεται εισρωή ατόμων, ε, όχι μόνο η γυρεότερη Ευρώπη, δηλαδή δεν είναι μόνο η γυρεά Ευρώπη που χρειάζεται αυτήν την ανανέωση εν ώψη ε, του, του δημογραφικού προβλήματος, των δημογραφικών τάσεων. Ε, Κατά τη γνώμη μου είναι εξοργιστικό ότι σε όλα τα μέτρα που έχουμε συζητήσει δεν αναφέρεται τίποτε για ε, τον άνοιγμα ε, νομίμων ε, διόδων και τρόπων ανθρώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας ε, ε, προσφύγων να μπορούν να ετούνται άσυλο όπως πρέπει και να μην χρειάζεται να περνάνε από λαθρέμπορους γιατί εμείς έτσι ενθαρρύνουμε τους λαθρέμπορους και αυτό είναι απαράδεκτο. Όταν ακούμε, όπως άκουσα προηγουμένως ε, στην Επιτροπή ε, ΛΥΜΠΕ, την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και Εσωτερικών Θεμάτων, μας είπε ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι α, είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί καταφέραμε να ε, εξαρθρώσουμε τις, τους λαθρεμπόρους, το δίκτυο λαθρεμπόρων, γιατί κάναμε μια συμφωνία με την Τουρκία. Ναι, αλλά ξέρετε, τώρα απλώς άλλαξαν διόδους. Περνάνε από την Αίγυπτο, περνάνε από την Αλβανία ε, έχουν απλώς μεταφερθεί. Ε, ξέρετε ότι αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους στη Μεσαιόγειο. Είναι γελίο λοιπόν να λέμε ότι δουλεύει η συμφωνία με την Τουρκία και γι' αυτό λύνεται το πρόβλημα ενώ οι άνθρωποι πηγαίνουν απλώς από άλλες οδούς. Ο ρόλος μας λοιπόν ως ε, ε, βουλευτών είναι πάρα πολύ σημαντικός να τονίσουμε όλα αυτά τα θέματα, να ρίξουμε φως σε όλη αυτήν την ε, συζήτηση δήθεν προσπάθειας αντιμετώπισης του προβλήματος του ε, προσφυγικού ε, και χρηματοδότησης των λύσεων. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει απαραίτητη ρύθμιση ώστε το κοινό σύστημα σύλλου να λειτουργήσει σωστά. Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Εμείς για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Κοινοβούλιο εδώ λέμε ότι το σύστημα αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Πρέπει όμως να έχουμε πραγματική αλληλεγγύη για να γίνει αυτό αυτό και πρέπει να ζητήσουμε αλληλεγγύη από τους ανθρώπους ε, που έρχονται να μας βρουν. Ήμασταν λοιπόν ε, ε, πολύ επικριτικοί έναντι των Αμερικανικών αρχών, μιλώντας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι ο θεματοφύλακας των συνθήκων, γιατί μας γιατί σε μια ε, χώρα σαν την Πορτογαλία, ε, γιατί στην ε, Ελλάδα, στο μη κυβερνητικό σύμφωνο δεν σεβόμαστε κάποια ποσοστά και υπάρχουν άλλες χώρες υπό την ηγεσία της Αυστρίας παραβιάζουν την συνθήκη του ΣΕΝ οι χώρες ε, Βίζεγκρατ παραβιάζουν τη συνθήκη ε, του ε, Σέγγεν και δεν γίνεται τίποτε. Δεν λέμε τίποτε για αυτές τις χώρες. Εγώ πραγματικά είμαι εξοργισμένη. Είμαι εξοργισμένη ότι τη στιγμή που η, Ουγγρα... Ουγγαρία άρχισε να χτίζει φράκτες ε, και να απορρίπτει κάτι το οποίο είχε ε, συμφωνηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν έγινε απολύτως τίποτε. Ε, και φυσικά οι χώρες Βίζεγκαρ μετά υπό την ηγεσία της Αυστρίας ε, και ενδεχομένως με τη χειραγώγηση άλλων κάποιον, ε, ενδεχομένω στη Γερμανία, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ε, η μεγάλη εισρωή είχε να κάνει με το γεγονός ότι πολλοί κόσμοι πίστευε ότι υπήρχε, ε, ένα, ότι υπήρχε μια θέση για εκείνους στη Γερμανία. Οι χώρες λοιπόν έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στην υποδοχή των ανθρώπων αυτών και μόνο να χειροκροτήσω μπορώ όσους το έκαναν αυτό όμως δυστυχώς ε, μετά άλλαξε η θέση ε, των χωρών αυτών ε, και δεν μπορώ να δω τι ακριβώς, ποιος ακριβώς είναι ο λόγος με αυτές τις χώρες Βίζεγκαρτ που ξαφνικά άρχισαν να χτίζουν φράχτες ή με την ε, επιβολή νομοθεσίας που είχε να κάνει με ε, τα ε, πυροβόλα όπλα. Έχω την εντύπωση ότι όλο αυτό είναι μια χειραγώγηση από κάποιους. Αποτυγχάνουμε κυρίες και κύριοι. Δεν ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας στο διεθνές δίκαιο και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των προσφύγων συνήφθη λόγω των Ευρωπαίων προσφύγων μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και συγκεκριμένα ε, Ούγγρων όχι μόνο βέβαια, μεταξύ άλλων. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που κάνουμε είναι ότι ουσιαστικά στρεφόμαστε ενάντια στη μας την, ε, στο δικό μας τον ανθρωπισμό, ε, στη δική μας την ιστορία. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχει προστασία των εξωτερικών συνόρων, αλλά δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει ακτοφυλακή ε, και με όλα αυτά που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται με παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των προσφύγων που έχουν τα δικαιώματα των πιο ευάλωτων, αυτών που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Πραγματικά είμαι εξοργισμένη. Πήγα στην Ιδωμένη, πήγα στην Ελλάδα. Ε, δεν υπάρχει μόνο μία Ιδωμένη τώρα, υπάρχουν χιλιάδες Ιδωμένες. Ε, οι άνθρωποι παραμένουν στην Ελλάδα, ε, μένουν σε αποθήκες, ε, σε τρομερές συνθήκες. είναι πραγματικά μία παγίδα θανάτου. Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης με τη ζώνη του Σέγγεν, γιατί η Ελλάδα δεν ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει αντιμετωπίζει μια τέτοια κατάσταση και ε, ε, δεν νομίζω ότι πραγματικά βοηθά κανείς όπως είχε υποσχεθεί την Ελλάδα πραγματικά γιατί ακόμη και με αυτή την διαδικασία ενσωμάτωσης που θα έπρεπε να λειτουργεί δεν λειτουργεί και ξέρω γιατί μιλάω γιατί έχω άμεσα συνεργαστεί με άλλους συνεδέλφους ε, με συγκεκριμένα 400 ανθρώπους που ήταν στην Ιδωμένη θα έπρεπε να έρθουν στην Πορτογαλία Τρει μήνε είναι εκεί και δεν έχει γίνει απολύτω τίποτα. Τίποτα απολύτω δεν γίνεται. Λοιπόν, συγγνώμη ε, που ε, σα ε, το λέω και σα το ξαναλέω, αλλά δεν πρέπει να ε, καταπίνουμε αμάσιτες ε, τις στρεβλές εικόνες που μας παρουσιάζονται. Ο ρόλος μας ως ε, βουλευτών είναι πάρα πολύ σημαντικός. Πρέπει να μιλούμε περισσότερο μεταξύ μας, να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και να δουλέψουμε γιατί πιστεύω και όλοι όσοι βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούν ε, σοβαρά να προσχωρήσουν, ε, είτε πιστεύουμε στις αξίες ε, και στις αρχές που διαμόρφωσαν αυτήν την Ευρώπη ή απλώς είναι μία λέσχη πλουσίων και τότε δεν είναι δική μου ένωση και δεν μπορεί να επιβιώσει. Δεν μπορεί να επιβιώσει γιατί δεν ε, υπάρχουν οχυρά, δεν υπάρχουν ε, ε, φράχτες που θα σταματήσουν τον κόσμο που έχει ανάγκη από το να προσπαθεί να έρθει. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γκομές για την παρέμβασή σας. Να δώσουμε το λόγο για ερωτήσεις, σχόλια, δηλώσεις, οτιδήποτε επιθυμείτε. Βλέπω πρώτο τον κύριο Γκέργεφ. Ευχαριστούμε κυρία Γκόμεσα. Δεν υπάρχει ΦΥΡΟΜ ως χώρα, δεν υπάρχει πουθενά. Η χώρα ονομάζεται Μακεδονία. Εγώ είμαι 37 ετών και έχω το δικαίωμα να αυτό προσδιορίζομαι και το ίδιο και οι ε, συμπατριώτες μου. Όλοι είναι Μακεδόνες. Όλοι είμαστε Μακεδόνες. Δεν υπάρχει ΦΥΡΟΜ εάν θέλετε να είστε υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του αυτοπροσδιορισμού της ελευθερίας έκφρασης, παρακαλώ σεβαστείτε το όνομα και τα συναισθήματά μας και την ταυτότητά μας, εμένα και της οικογένειάς μου. Δεν θα πάθετε τίποτα αν πείτε ότι είμαστε Μακεδόνες, είμαι Μακεδόνας και παρακαλώ να μου απευθύνεστε ως Μακεδόνα και στη χώρα μου ως Μακεδονία. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ηλιάνης, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμα μέλη, θα ήθελα να σχολιάσω το πρώτο κομμάτι της παρουσίασής σας Είμαι μέλος της αντιπολίτευσης του Κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου και είμαι μέλος της Επιτροπής ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ελευθεριών και είμαι πρώην μέλος ε, της Επιτροπής για Αμυντικά Θέματα και Θέματα Ασφαλείας. Θα ήθελα να σχολιάσω για το πρώτο κομμάτι της ομιλίας της κυρίας Γκόμες ε, που αφορά τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια. Όπως ακούσαμε, οι πρόσφυγες δεν αποτελούν την κύρια απειλή προς την ασφάλεια και συμφωνώ με αυτό. Οι αλλοδαποί μαχητές ε, ουσιαστικά είναι υπήκοοι των δικών μας χωρών που μεταβαίνουν σε χώρες ε, σειράξεων στο εξωτερικό και επιστρέφουν και αυτή είναι η μεγαλύτερη απειλή. Συμφωνώ με αυτό και εγώ ως βουλευτής του δικού μου κοινοβουλίου ήμουν από τους πρώτους στα Βαλκάνια που ανέλαβε την πρωτοβουλία να αλλάξει τον ποινικό κώδικα του Μαυροβουνίου, πράγμα που συνέβη. Αλλάξαμε τον ποινικό κώδικα, τον βελτιώσαμε θα έλεγα, ώστε το... οι υπήκοοι του Μαυροβουνίου που μεταβαίνουν σε χώρες Ιράξεων, στο εξωτερικό, ε, τιμωρούνται με φυλάκιση. Άμα επιστρέψουν. Και με κάποιο τρόπο έτσι συμβάλαμε στην όλη προσπάθεια. Αλλά φυσικά δεν αποκλείω αυτό τον κίνδυνο της τρομοκρατίας. Δεν τον συζητήσαμε εκτενώς βέβαια εδώ. δεν χρειάζονται πολλοί πρόσφυγες ε, που να θέλουν να εμπλακούν σε τρομοκρατικές ε, δράσεις. Χρειάζονται ελάχιστοι για να βλάψουν αθώους ανθρώπους. Και όπως οποιαδήποτε χώρα στην Ευρώπη ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε σοβαρές καταστροφές με πολλά θύματα. Και αυτή, αυτό είναι ένα ενδεχόμενο διότι από τα εκατομμύρια των προσφύγων είναι απίθανο να μην υπάρχει κανένας που να έρχεται με άλλες προθέσεις της χώρας μας. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Με αυτή την ε, νοτροπία καταστροφής. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειαζόμαστε στενή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμάς που φιλοδοξούμε να προσχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να ανταλλάσσουμε δεδομένα και να έχουμε στενή συνεργασία. Θα έλεγα επίσης και συνεργασία μεταξύ κοινοβουλίων, κοινοβουλευτικών οργάνων και των εκτελεστικών εξουσιών, των υπηρεσιών ασφαλείας, των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, των αστυνομικών αρχών και ούτω ώστε να αποφύγουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είναι πολύ αργά πια για να τα συζητήσουμε. Διότι αφού συμβούν τέτοια περιστατικά, είναι πολύ, πια, πολύ αργά πια για να τα συζητήσει κανείς. Το έχουμε ξαναβιώσει στο παρελθόν. Δεν θέλουμε να επαναληφθούν τα ίδια. Αρκεί μία περίπτωση τέτοια για να στιγματιστούν, στιγματίζονται όλοι οι μετανάστες ως τρομοκράτες. Και αυτό αποτελεί επιπλέον φόρτο τόσο για αυτούς όσο και για εμάς όπου βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου καλούνται να αιτιολογήσουν κάτι το οποίο είναι δύνατο να αιτιολογηθεί. Χρειαζόμαστε πιστεύω λοιπόν να παρακολουθούμε στενά τα όσα συμβαίνουν όλοι μας από κοινού και συνεργαζόμενοι. Και μέσω αυτής της συνεργασίας μεταξύ όλων των αρμόδιων φορέων να προλάβουμε τέτοια περιστατικά. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να σχολιάσω. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις χώρες, στη Συρία, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ. Οι περισσότεροι πρόσφυγες έρχονται από αυτές τις χώρες. Φαντάζομαι ότι αν θέλετε να αντιμετωπίσετε το ζήτημα, το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να αντιμετωπίσετε τα αίτια και τα αιτία κρύβονται φανταζόμενες στις χώρες καταγωγής αυτών των προσφύγων. Σε τέτοιες ε, συνθήκες κρίσης θα έλεγα ότι όλοι μας στα Δυτικά Βαλκάνια έχουμε βιώσει αυτή την τραυματική εμπειρία των σειράξεων και των μεταναστών. Το 20% των κατοίκων του Μαυροβουνίου κάποια στιγμή ήταν ε, μετανάστες. Το έχουμε ζήσει δηλαδή και ρωτάω, έχει μηχανισμούς η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναλαμβάνει δράσεις στις χώρες καταγωγής αυτών των ε, προσφύγων. ώστε να προσπαθήσει να διορθώσει κάποια πράγματα εκεί, ώστε οι άνθρωποι να μένουν στις χώρες τους, στα σπίτια τους. αποφεύγοντας ε, αυτό, το επικίνδυνο εγχείρημα της μετανάστευσης. Ακούμε ότι πολλοί από αυτούς ε, έχασαν μάλιστα τραγικά τη ζωή τους στη διαδρομή αυτή. Ευχαριστούμε κύριε Μερένιτς. Ο επόμενος ομιλητής η κυρία Καρακώστα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η αλήθεια είναι ότι <clears throat> στη σημερινή σύσκεψη δεν θα ήθελα να μπει το θέμα ε, που μπήκε σε σχέση με την ονομασία Φύρομ Είμαι όμως αναγκασμένη να τοποθετηθώ σε αυτό και να πω ότι αντιλαμβάνομαι τους ανθρώπους που λένε ότι γεννήθηκαν πιστεύοντας ένα όνομα. Αν όμως πάρω αυτό το κριτήριο, ξέρετε, εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερη σας και σας θυμάμαι ως Ιγκοσλαβία. Ε, άρα λοιπόν ε, να μπούμε στα νέα δεδομένα, να λάβουμε την επίσημη αποδοχή της ονομοσίας Φύρο αυτή τη στιγμή και ας μπει σε άλλες συσκέψεις ή οποιοδήποτε αίτημα ε, φαντάζομαι από την πλευρά των ε, Σκοπίων. Και αυτό γιατί, γιατί σήμερα βρισκόμαστε σε μία σύσκεψη που προσπαθούμε να ενοποιήσουμε τις απόψεις μας σε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και είναι κρίμα να βρίσκουμε τις διαφορές αντί τα στοιχεία ενότητάς μας. Επίσης, θα ήθελα σχετικά με αυτό που είπε ο συνάδελφος από το Μαυροβούνιο που συνέδεσε την τρομοκρατία με το προσφυγικό, πραγματικά επίσης δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Δεν πρέπει δηλαδή να βρούμε τον έναν που ψάχνει, πιθανά κάποιος από φόβο να βρει ως πέρασμα, και αυτό να το συνδέουμε με το σύνολο των προσφύγων. Ε, το προσφυγικό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και δεν πρέπει να ξεχάσουν αυτές οι χώρες που προέρχονται από την πρώην Ιουγκοσλαβία πως η Ελλάδα δέχτηκε πάρα πολλούς πρόσφυγες από την πλευρά ε, αυτής της διάσπασης της, αυτής της χώρας. Όπως επίσης δέχτηκε εξαιρετικά πολλούς πρόσφυγες, οικονομικούς μετανάστες από την Αλβανία, από τη Βουλγαρία, από τις χώρες του πρώην σοσιαλισμού. Άρα λοιπόν αυτή η μετακίνηση των πληθυσμών, είτε είναι πρόσφυγες πολέμου, είτε είναι πρόσφυγες οικονομικοί μετανάστες, πρέπει να το δούμε στα πλαίσια που εξαιρετικά έβαλε η κυρία Γκομές. Ε, έτσι οφείλουμε να το δούμε, διότι είμαστε χώρες που ειλικρινά δημιουργήσαμε νέες χώρες από την Επανάσταση, από την, από την προσφυγιά, συγγνώμη. Μην ξεχνάτε ότι ε, στην πλειοψηφία της η Αμερική είναι οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι. Ε, μην ξεχνάμε όλο αυτό. Μην ξεχνάμε ότι ελληνισμό έχουμε στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Αμερική, πέρα από τις χώρες της Ευρώπης. Είμαστε λοιπόν όλοι άνθρωποι που προέρχονται και γεννήθηκαν σε διαφορετικές χώρες, άλλοι βρίσκονται στις χώρες, σε άλλες χώρες. Έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως κίνηση πληθυσμών. Και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα, βεβαίως μη δημιουργώντας πολέμους σε αυτές τις χώρες που σήμερα έχουν πόλεμο, μην εκμεταλλευόμενοι τις πλουτοπαραγωγικές πηγές χωρών που δεν βρίσκονται οικονομικά και τεχνολογικά αναπτυγμένες, πηγαίνοντας εμείς, παίρνοντας τον πλούτο, φέρνοντάς τον στις χώρες μας, αφήνοντάς τους φτωχούς και μετά λέμε οικονομικοί μετανάστες. Άρα λοιπόν ένα γενικότερο σύνολο πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας, αν πραγματικά θέλουμε να είμαστε η Ευρώπη εκείνων των ιδεών της ελεγγύης, εκείνων των ιδεών της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και πολλών άλλων ε, ωραίων τίτλων. Αυτά θα ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, madam. Yes, please. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ονομάζομαι Νάντζα Τσιμπούσεβα από το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Και θέλω πολύ σύντομα να απευθύνω χαιρετισμό Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές χρήσιμες συζητήσεις, επικοδομητικές, πολλά θέματα συζητήθηκαν. θα έγινε λόγος για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις, ε, στην προσπάθειά τους για μετανάστευση η μετανάστες. Θα ήθελα να αναφερθώ στα όσα είπε η συνάλφος από την νότια γείτονα, την Ελλάδα. Είμαστε η Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτό είναι το νόμιμο δικαίωμα, το ανθρώπινο δικαίωμά μας. Και έχουμε δικαίωμα να αποκαλούμεθα Δημοκρατία της Μακεδονίας, γιατί είμαστε Δημοκρατία της Μακεδονίας και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Ας αφήσουμε όμως τα νομικά ζητήματα. Έχουμε άλλα θέματα να συζητήσουμε. Γι' αυτά ήρθαμε εδώ. Έχουμε να κάνουμε με τη μεταναστευτική κρίση όπου και Μακεδονιακές μην είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πλάκη. Υπάρχει μια γεωστρατηγική θέση, η οποία μας έφερε πάνω στο δρόμο της μετανάστευσης. Η Δημοκρατία της Μακεδονίας ήταν πύλη υποδοχής προσφύγων από μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης περνούσαν για να πάνε σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημοκρατία της Μακεδονίας έχει διδραματίσει σημαντικό ρόλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ας αναφέρθηκε ότι κλείνουμε σύνορα. Δεν τα κλείσαμε εμείς τα σύνορα όμως. Μόνοι μας. Κλείσανε με βάση τους κανόνες που επέβαλαν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι βόρειοι γειτονές μας. Εκείνοι που έφραξαν τους δρόμους της μετανάστευσης. Και έτσι κατέστησαν για μας αδύνατο να υποδεχθούμε τους μετανάστες και να εξασφαλίσουμε την περαιτέρω μετάβασή τους σε άλλες χώρες. Είμαστε μικρή χώρα Η δυνατότητα λοιπόν για υποδοχή μεταναστών που έχουμε, που διαθέτουμε είναι περιορισμένη. Και βέβαια χρειαζόμαστε οικονομικούς πόρους. Δεν έχουμε ως χώρα τέτοιες δυνατότητες εμείς. Νομίζω ότι έχουμε αντιμετωπίσει με πολύ ικανοποιητικό τρόπο τη μεταναστευτική κρίση και έχουμε βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση Είμαστε λοιπόν η Δημοκρατία της Μακεδονίας, είμαστε Μακεδόνας, πρόκειται για συνταγματικό και ανθρώπινο δικαίωμα και αυτό είναι το, το όνομα που θα χρησιμοποιούμε. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητεί κανείς άλλο το λόγο και τελειώνει και ο χρόνος. Ας παρακαλέσω λοιπόν την κυρία Γκόμες να δώσει απαντήσεις. Χωρίς μικρόφωνο. Χωρίς μικρόφωνο η κυρία Γκόμες. Η κυρία Γκόμες δεν ακούγεται. Ε, θα ζητήσω συγγνώμη και κατανόηση από την αντιπροσωπεία της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Θα εξακολουθήσω να χρησιμοποιώ το όνομα αυτό και το ακρονίμιο αυτό χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν, απλώς για να μην φέρω στη συζήτηση ακριβώς αυτή τη διαμάχη που εξακολουθεί να υπάρχει. Αυτό είναι το επίσημο όνομα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό χρησιμοποιούμε. Μακεδονία υπάρχει, υπάρχει και πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία. Αυτό δεν ήθελα. Το θέμα αυτό. Να μείνει εκκρεμές, θα ήθελα να επιληθεί βεβαίως με βάση τα δικαιώματα των πολιτών. Και θα ήθελα να πω ότι είμαι ευγνώμων για τα όσα είπατε, κυρία συνάδελφε. Αυτό ήταν και ο λόγος για τον οποίο διατύπωσα τις ερωτήσεις μου τις προάλλες. Ε, είπατε βεβαίως ότι η χώρα σας είναι μικρή, έχει περιορισμένους πόρους, βεβαίως, όπως και η δική μας χώρα. Και ότι υπάρχουν ε, πολλές πιέσεις. πιέσεις σε σχέση με τους γείτονες, πιέσεις όταν κανείς βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Αλλά πολύ σωστά λέτε ότι όταν υπάρχει απόφαση για παραβίαση της Συμφωνίας Σέγγεν από κράτη-μέλη, θα πρέπει βεβαίως να φέρουν και τη σχετική ευθύνη κυρίως όταν αυτή η απόφασή τους επηρεάζει και άλλα κράτη. Για τον κύριο Μίλανιτς από την αντιπροσωπεία του Μαυροβουνίου. Συμφωνώ βεβαίως με τα όσα είπατε, Αφελή δεν είμαι. Ένα μέρο τη δουλειά μου σχετίζεται στενά με την καταπολέμηση τη δημοκρατίας. Βεβαίω και ξέρω ότι είναι οπορτινιστέ οι τρομοκράτε και θα αξιοποιήσουν κάθε δυνατή ευκαιρία. Ταυτόχρονα όμως αυτοί οι άνθρωποι που προσπαθούν να ξεφύγουν από το Ιράκ, τη Συρία, από τον πόλεμο και την τρομοκρατία προσπαθούν ε, να ξεφύγουν. Το Ιράκ το επισκέφθηκε πριν από ένα χρόνο ανάμεσα στις επιθέσεις κατά του ε, Σαρλί την πρώτη και μετά του Μπατακλάν. Και ήρθαν οι Ιρακινοί όταν τους συνάντησα και μου είπανε όλοι αυτοί, αυτοί οι οποίοι ε, δίωκαν και ε, έσφαζαν τους Γεζιδί και τους Χριστιανούς και όλους αυτούς. Είναι Ευρωπαίοι. Είναι οι δικοί σας τρομοκράτες. Και στο Ιράκ που πήγα και επισκέφθηκα καταβλισμούς, όλοι μου λέγαν ότι με την πρώτη ευκαιρία θα ερχόντουσαν στην Ευρώπη. Γιατί μπορεί να υπήρχαν καταβλισμοί, αλλά εκπαίδευση δεν είχαν δυνατότητα να εξασφαλίσουν για τα παιδιά τους. Πολλοί λοιπόν λέγανε ότι θα έρθουν τουλάχιστον για να έχουν τα παιδιά τους μια ευκαιρία στην εκπαίδευση. Ναι λοιπόν, έχουμε τεράστιε ευθύνε. Μεγάλο μερίδιο τη ευθύνη. Όχι ολόκληρη βέβαια. Και αν κοιτάξει και κανεί πώ διανέμεται η ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι γελία η κατάσταση. Την εκπαίδευση την έχουν τελείως παραγνωρίσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτό ήταν και ένα λόγο από τον οποίο οι άνθρωποι εξαναγκάστηκαν να φύγουν. Μέσω τη Τουρκία βεβαίω πολύ. Αλλά πάντα μας έχουν την Ευρώπη. Και δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι δεν το ήξερε. Από εδώ. Το ξέραμε πολύ καλά. Και εγώ το έλεγα πάντα ότι θα συμβεί αυτό. Γιατί είχα επισκεφθεί αυτές τις χώρες, είχα δει με τα μάτια μου. Έχουμε πολλές αντιπροσωπείες ε, και στην Ιορδανία και στον Λίβανο. Που είδαμε μια απίθανα γενναιόδορη προσέγγιση απέναντι στους πρόσφυγες. Με, όλο το, με όλη την επιβάρυνση και την πίεση που σημαίνει για τον πληθυσμό του. Πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθούμε και νομίζω ότι αυτό δεν έχει εξασφαλιστεί. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν είναι γελίο να περιγράφονται ως τρομοκράτες. Προσπαθούν να ξεφύσουν από τους τρομοκράτες και από τον πόλεμο. Τρομοκράτες υπάρχουν φυσικά, αλλά είναι εδώ, μεταξύ μας. Το να λέμε τους ε, ανθρώπους αυτούς, ε, τους πρόσφυγες τρομοκράτες, όπως κάνει άκρα δεξιά, εξυπηρετεί ακριβώς το παιχνίδι των ίδιων των τρομοκρατών του ίσης. Ξέρουμε παραδείγματι ότι έχουν ε, χρησιμοποιήσει ε, διαβατήρια ε, τότε με την επιθέση του Μπατακλάν στη Γαλλία. Ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί θέλανε τον μετανάστη εμείς να τον δούμε σαν υποψήφιο τρομοκράτη. Γιατί αυτό θέλανε. Ας είμαστε λοιπόν ευφιέστεροι αυτού. Πόσους ανθρώπους δεν μετατρέπουμε σε πιθανούς εξτρεμιστές σε ανθρώπους που μισούν τις κοινωνίες μας. Εάν τους αφήνουμε αβοήθειο, αβοήθητους χωρίς καμία ενσωμάτωση κοινωνική. Οι ανήλικοι. Πάνω από 10.000 ανήλικοι λέγεται πως έχουν εξαφανιστεί ενώ έχουν φτάσει στα εδάφη των ευρωπαϊκών κρατών. Πού είναι τα παιδιά αυτά. Πού είναι αυτοί οι ανήλικοι. Κάποια από αυτά τα παιδιά μπορεί ήδη να έχουν πέσει θύματα ε, δικτύων ε, είτε για σεξουαλική εκμετάλλευση, είτε για ε, όργανα προς μεταμόσχευση. Πολλά από αυτά μπορεί να ξεφύγουν μεν, αλλά χωρίς καμία δυνατότητα για κοινωνική ενσωμάτωση. Για σκεφτείτε όλοι αυτοί, όλα αυτά τα παιδιά τι δυναμικό για τρομοκρατία μπορεί να εκπροσωπούν για το μέλλον. Το δικό μας συμφέρον κοιτάμε, το δικό μας συμφέρον υπερασπιζόμαστε. Πρέπει λοιπόν και αυτό να το κοιτάξουμε. Δεν πρέπει να το αγνοήσουμε το πρόβλημα. Είναι παντού όμως. Για δείτε οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πόσο φασαρία κάναν για το PNR, το σύστημα καταγραφής στοιχείων επιβατών πτήσεων για να βρίσκουν τους τρομοκρατές. Αλλά υπάρχει το παραθυράκι. Οι ιδιωτικές πτήσεις. Γιατί μπορεί ωραιότατα ένας τρομοκράτης να νοικιάσει ιδιωτικό ε, αεροπλάνο και να έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να καταγραφούν τα στοιχεία του που θα... Να, δεν τον δυσκολεύει σε αυτό κανείς. Ξέρουμε ότι εμείς σε μεγάλο βαθμό έχουμε διευκολύνει τους τρομοκράτες και την παρουσία τους εδώ. Αλλά πρέπει να είμαστε βέβαια προσεκτικοί. Και γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε αποτελεσματικές διαδικασίες ε, ε, επιτήρησης, παρακολούθησης, ελέγχου των εξωτερικών συνόρων, αποτελεσματική συνεργασία με τους λοιπούς εταίρους που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα γειτονικά κράτη κτλ. Όλα δυστυχώς αυτά είναι διάτρητα, είναι γεμάτα παραθυράκια. Δεν εξασφαλίζουν τους όρους ασφαλείας που απαιτούνται. Και βέβαια ξέρω ότι είναι τεράστιος ο φόρτος, τεράστια επιβάρυνση για τις χώρες που έρχονται με αυτές τις τεράστιες ροές. Δεν πρόκειται όμως να εξαφανιστούν, δεν πρόκειται να πάψουν αυτές. Θα σταματήσει ο ένας πόλεμος, θα αρχίσει ο άλλος. Το θέμα λοιπόν είναι ότι χρειαζόμαστε πολιτικέ, ε, ολοκληρωμένες πολιτικές και εξωτερική πολιτική με διάσταση επίλυση κρίσεων, συγκρούσεων και πάνω απ' όλα πρέπει να διορθώσουμε όλα αυτά τα τεράστια λάθη που έχουν γίνει στο παρελθόν και που δεν βοηθούν να μειωθούν οι ροές. Αντιθέτως, όλο και μεγαλύτερες είναι οι ροές. Επιμένω. θα έπρεπε να αναφέρουμε όντως ε, νομότυπους και ασφαλείς τρόπους. Έτσι το κλείνουμε το μαγαζί του λαθρομδιακινητή. Αλλά είναι δυστυχώς πολύ στενόμελη η προσέγγιση των κρατών, των κυβερνήσεων. Και δεν το έχουν δεχθεί μέχρι τώρα. Ένα άλλο μέσο που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε, αλλά δεν υπάρχει ακόμα, θα ήταν μια προσωρινή ε, προστασία ασύλου. Κάτι που είχε εφευρεθεί την εποχή του λέμε, της Ιουκοσλαβίας και θα μπορούσαν τα κράτη μας να το αξιοποιήσουν για να προσφέρουν την προστασία σε εκείνους που την ε, χρειάζονται και που θα είναι έτοιμοι μετά να γυρίσουν στις πατρίδες τους όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες. Ε, νομίζω ότι από τους πρόσφυγες, από όλους αυτούς τους πρόσφυγες με τους οποίους έχω συνομιλήσει, είναι σαφές ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν αφήσει τη χώρα τους, την πατρίδα τους, γιατί τους αρέσουν τα ταξίδια. Αναγκάζονται να φύγουν γιατί είναι διοκόμενοι, γιατί κινδυνεύουν, κινδυνεύει η ζωή τους. Θέλουν να γυρίσουν στις πατρίδες τους. Και σε αυτό πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε, να τους ενσωματώσουμε στο δυνατόν περισσότερο και βέβαια να τους βοηθήσουμε να επιστρέψουν στις πατρίδες τους και να τους βοηθήσουμε να ανεκοδομήσουν τις πατρίδες τους. Με λύπη μου θα πω ότι δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα. Και αυτό καθήκον θα πρέπει να το παραδώσουμε στις επόμενες γενναίες μακροπρόθεσμα όλο και περισσότερο θα πρέπει τα κοινοβούλια να κοιτούν και να εξετάζουν τι κάνουν οι κυβερνήσεις μας, τι κάνουν οι ε, δομές οι κρατικές. Να μην εγκαταλείπουμε τους ανθρώπους αυτούς. Γιατί δεν νομίζω ότι έτσι εξυπηρετούμε κανέναν και πάντως όχι της κοινωνίας μας. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας και για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κόμες και έτσι φτάσουμε στο τέλος ε, της ε, διάσκεψής μας. Τις δύο αυτές μέρες συζητήσαμε για το ρόλο των κοινοβουλίων ε, όσον αφορά την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης. Μιλήσαμε για την αντιμετώπιση τη τρέχουσα κρίση ε, με υπευθυνότητα και με ένα μηχανισμό αλληλεγγύη. Ακούσαμε διάφορε παρουσιάσει ε, για το ρόλο των κοινοβουλίων ε, στο να παρέχουν απόκριση στα διάφορα ζητήματα της διαχείρισης συνόρων, τη μετανάστευση του ασύλου. Σήμερα ακούσαμε ακόμη περισσότερα για την κατάσταση στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους ρόλους των κοινοβουλίων στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων και στη διαχείριση των κρίσεων. Ελπίζω ειλικρινά να βγείτε από αυτή την αίθουσα με κάποια έμπνευση, κάποιες νέες ιδέες ε, και με κίνητρα για να συνεχίσετε τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαχείριση ε, μίας από τις εντονότερες κρίσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα. Το πρόβλημα είναι τεράστιο, είναι αδύνατο να το επιλύσουμε με μία διάσκεψη, αλλά πιστεύω ότι ήταν καλό που ανταλλάξαμε απόψεις και θέσεις για το τι προσέγγιση θα πρέπει να ακολουθήσουμε για αυτό το θέμα στο μέλλον. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σας. Ήταν μεγάλη μας χαρά να σας έχουμε εδώ και παρότι ήταν μικρό το διάστημα που εγώ πρόεδρεσα ε, αυτή τη συνεδρία. μου ήταν πολύ ευχαριστώ να σας ευχηθώ καλή επιστροφή στα σπίτια σας και Εύχομαι να είναι θετικέ και αποτελεσματικέ ε, οι μελλοντικέ σα δραστηριότητε στην πολιτική σα ζωή. Ευχαριστώ. Κύριε Σωτοπέρα, συνειδητή.